So good morning everybody, welcoming those who are here in time. Καλημέρα, λοιπόν. Κάποιοι έχουν έρθει στην ώρα τους, αν και έχουμε καθυστερήσει ήδη λίγο, αλλά έτσι θα έχουν και άλλοι συνάδελφοί την ευκαιρία να φτάσουν. Πρώτο θέμα, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει καμία παρατήρηση, όχι, εγκρίνεται. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Έχω αρκετές, με συγχωρείτε. Λοιπόν, IORP έγινε πολύ καλή πρόοδος στο διάλογο της 5ης Ιουνίου, πήγαμε μετά τα μεσάνυχτα, οπότε κάτι κάναμε ειδικά. Πρόοδος σημειώθηκε για τις διασυνοριακές δραστηριότητες, όπου τώρα αναγνωρίζαμε πως μπορεί να υπάρξει μια υποχρηματοδότηση όταν υπάρχουν διασυνοριακές συναλλαγές και άρα θα πρέπει να ληφθεί ανάλογη δράση για να επανέλθει η κατάσταση στο φυσιολογικό. Διασυνοριακή μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όπου θα υπάρχει μια πρώτερη εξοδότηση του κράτους μέλους όπου ε, υπάρχει αυτή η μεταφορά. Στην ε, δε περίπτωση και του κράτους ε, προορισμού το ίδιο. Στην ε, ισορροπία μεταξύ των γενεών θα πρέπει να υπάρξει ένας ίσως καταμερισμός ε, των κινδύνων και του ωφέλους μεταξύ των γενεών. Περιβαλλοντική διακυβέρνηση θα πρέπει να εξετάζονται και οι σχετικοί κινδυνοί όταν λαμβάνονται οι σχετικές επενδυτικές αποφάσεις καθώς μπορεί τώρα να έχουν υψηλές αποδόσεις οι εταιρείε αλλά όχι στο μέλλον. Μετά έχουμε μια δήλωση συνταξιοδοτικών ε, δικαιωμάτων όπου αντί για πλήρως εναρμονισμένη έχει, έχουμε πάει σε μια δήλωση που θα βασίζεται σε αρχές και βασιζόμαστε εδώ πέρα στην γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης. Αυτά λοιπόν για τα συνταξιδοτικά ταμεία. Η Εξεταστική Επιτροπή, ναι, λοιπόν, έχουμε την τρίτη οδηγία για τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπου ξεκαθαρίζουμε ότι διατάξεις ε, περί επαγγελματικού απορρίτου, ελπίζω να μην σας ενοχλώ, Ε, επειδή μιλάμε για επαγγελματικό απόρριτο, ισχύουν χωρίς να επηρεάζουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 226 της συνθήκης. Υπάρχουν ορισμένα εκρεμή ζητήματα πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία και αναμένουμε ότι αυτό θα συμβεί πριν το τέλος Ιουνίου. Ελπίζουμε λοιπόν η Ολλανδική Προεδρία να καταφέρει να κλείσει το θέμα και χάρη στην δική μας διαπραγματευτική ομάδα. Για τη σημερινή συνεδρίαση υπενθυμίζουμε πως θα λάβει η χώρα μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΕΜΠΛ σήμερα και βεβαίως θα ξαναλλάξουν μετά τα έδρανα για την απογευματινή συνεδρίαση που θα έρθει ο κύριος Δράγκης. Μπορούμε άρα τώρα να περάσουμε σε κάποιες πληροφορίες για την τελευταία συνεδρία των συντονιστών 15 Ιουνίου. Σύνοψη συστάσεων και αποφάσεων. Ορίσμη λάβαμε την έκθεση για την τέταρτη οδηγία κατά του ξεπλήματο χρήματο Από κοινού με την Επιτροπή Λίμπε που θα πάει... Αυτή πάει στο ΕΛΚ. Πρόγραμμα της Ένωσης για στήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για τελικού χρήστε στον καθορισμό της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής, πάει πράσινες βεβαίως, αποκάλυψη πληροφοριών φόρου εισοδήματος από κάποιες επιχειρήσεις. Ζητήσαμε να εφαρμοστεί το άρθρο 55 να είμαστε κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή, πάει σοσιαλδημοκράτες, ε, τραπεζική ένωση ΕΛΚ, FinTech, ό,τι και αν σημαίνει αυτό στους φιλελεύθερους. Α, το ξέρετε εσείς τι σημαίνει, ωραία. Γιατί εντάξει, αυτό σημαίνει τα πάντα και τίποτα. Λειτουργία τη δικαιώχησης στον τομέα τη Λιανική. γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 54, Σοσιαλδημοκράτε. Ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ο Πρόεδρος θα απευθύνει επιστολή στην διάσκεψη των Πρόεδρων Επιτροπών για να συντάξουμε δύο σχέδια έκθεσης για την IGS και τις συστάσεις της Ευρωζώνης με στόχο της Ολομέλειας Φεβρουαρίου και Οκτωβρίου του 2017. Θα απευθύνουμε επιστολή στον Πρόεδρο για να ζητήσουμε να ξεκινήσει άμεσα η εργασία η οποία αναφέρεται στην έκθεση των πέντε Πρόεδρων για την Ομάδα Εργασίας Οικονομικής Βοήθειας. Είχαμε την ενημέρωση με τα θεσμικά όργανα η οποία πρέπει να προσθεθεί στο πρόγραμμα. Ακρόαση με την ΕΚΤ, την Επιτροπή Προσωπικού και τα Συνδικάτα θα οργανωθούν δύο διαφορετικές ε, ακροάσεις, μία με την ΕΚΤ και η δεύτερη κατά προτίμηση αμέσως μετά για να δούμε την άποψη των εργοδοτών. Ε, οικονομικός διάλογος με κράτη-μέλη υπάρχουν τρεις εκρεμείς προσκλήσει ε, που είχαμε απευθύνει το 2015 σε Κροατία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ζητήθηκε αυτή η γραμματεία να τις ε, παρακολουθήσει, να δει τι γίνεται και θα ακολουθήσει η Ισπανία και η Πορτογαλία μετά τις διακοπές. Εξέταση πράξεων κατεξιοδότηση. Θα έχουμε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα στις 16 Ιουλίου το θέμα για την 31 Σεπτεμβρίου, 1η Οκτωβρίου, η οδηγία για την φερικαιότητα 2 και ελπίζω να μην γίνει μη Διεθνή λογιστικά πρότυπα 9. Συντονιστές ε, ενέκριναν μια επιστολή στον Επίτροπο για να αναφερθούν διάφορες ανησυχίες όσον αφορά την έγκριση του Διεθνών Λογιστικών Πρωτοβουλίων 9. Επίσης, οι συντονιστές συζήτησαν τη διαδικασία έγκρισης εν ώψη των διακοπών και συμφώνησαν πως η ψηφοφορία θα πρέπει να λάβει χώρα στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 και μετά να πάει στην Ολομέλεια την 1η του Οκτωβρίου. Μελέτη του ανταγωνισμού εγκρίναμε μία πρόταση να αναθέσουμε μία μελέτη που θα μας δώσει μία γενική εικόνα για το πώς μπορούν να συνεισφέρουν τα μέσα που έχει Κομισιόν στην διάθεσή της για να επιτύχουμε μια εσωτερική αγορά ενέργειας, για να υπάρξει μια ενεργειακή ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιπρόσθετες ανακοινώσεις μετά από τα όσα μας είπε ο εισηγητής, συμφωνήσαμε να διατηρηθεί η ψηφοφορία για την έκθεση ΦΠΑ στις 13 Ιουλίου και να γίνει μια ακρόαση μετά τις διακοπές αλλά πριν την Ολομέλεια. Λοιπόν, ψηφοφορία, ακρόαση, Ολομέλεια με αυτή τη σειρά δια... κοινοβουλευτική διάσκεψη για την οικονομική διακυβέρνηση και τη σταθερότητα στην Πρατισλάβα για να μην συμπέσει αποφασίστηκε να ακυρωθεί η συνεδρίασή μας για τις 17 Οκτωβρίου και να ψάξουμε άλλη ημερομηνία για τη δημόσια ακρόαση. Συνεδρίαση της Επιτροπής Δευτέρα 27 Ιουνίου συμφωνήσαμε να γίνει από τις 3.30 μέχρι τις 7.30 το απόγευμα. Αυτά από ανακοινώσεις. Περνάμε τώρα στον έλεγχο εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών μέτρων. Και θα έχουμε τώρα την συζήτηση για τον κανονισμό για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Δίνω τον λόγο στον ε, εισηγητή, ο οποίος θα συνεχίσει τα γερμανικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα να δώσω τον λόγο στον κύριο Λούιντε από την Γενική Διεύθυνση Φύσμα και τον Στίβεν Μαγιόρ από την ΕΣΜΑ. Να με συγχωρείτε. Όχι, όχι. Λοιπόν, χαίρομαι που ήρθατε ξανά εδώ για να συζητήσουμε για το ΜΥΦΙΔ και το ΜΥΦΙΡ. Έχουμε προβλέψει πέντε λεπτά για τον καθένα, τα εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές και αν υπάρχει χρόνος και τσιάει. Για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, δίνω τον λόγο στον κύριο Στίβεν Μαγιόρ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Μάρκους, που μου δίνεις το λόγο και όντως ε, είναι πολύ σημαντικό να καλύψουμε και αυτή την ε, τελευταία συνεδρίαση ελέγχου όσον αφορά το MIFID. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσω μαζί σας με τα μέλη τη Επιτροπή Οικονομική Πολιτική για το πώ εφαρμόζεται οδηγία για τι αγορέ χρηματοπιστωτικών μέσων. Η εφαρμογή αυτή είναι πολύ σημαντική προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι στόχοι τη MIFID 2 που έχουν θέσει οι συνομοθέτε όντω επιτυχάνονται στην πράξη. Η ΕΣΜΑ υπέβαλε 42 σχέδια τεχνικών προτύπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το MIFID 2 και το MIFIR το 2015 αφού ολοκλήρωσε τη διαδικασία τεχνικής παροχής ε, συμβουλών το Δεκέμβριο του 2014. Για τρία από τα σχέδια αυτά προτύπων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε στην ΕΣΠΑ ότι θέλει να επιφέρει τροποποίηση, που σημαίνει ότι η ΕΣΠΑ περιμένει ότι η πλειονότητα των προτύπων τελικά εν ευθέτω χρόνο θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρί τροποποίηση. Όσον αφορά τις προσφάτως εγκριθήσεις εξώτηση πράξη, με χαρά βλέπω ότι όσον αφορά την προστασία των επενδυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τις τεχνικές συμβουλές της ΕΣΜΑ του ε, Δεκεμβρίου 2014. Η ΕΣΜΑ έχει επίση εκπονήσει τρει γνωμοδοτήσει για τα πρότυπα εκείνα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα έχει πει ότι θέλει να τα εγκρίνει μέσω τροποποιήσεων, ενώ συμφωνεί με τη γενικότερη προσέγγιση τη ΕΣΜΑ. Αυτά έχουν να κάνουν τα θέματα τη διαφάνεια για τα μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα, τα όρια θέσεων και τι παρεπόμενε δραστηριότητε. Και τα τρία αυτά θέματα είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστούν, ενώ θα πρέπει να σεβαστούμε και το κείμενο του πρώτου επίπεδου της ΜΥΦΙΤ 2 και να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για τις επιστολές της 27ης Νοεμβρίου του 2015 και της 7ης Απριλίου του 2016 για τα πρότυπα αυτά. Έχουμε λάβει υπόψη το περιεχόμενο των επιστολών αυτών κατά την κατάρτιση των γνωμοδοτήσεών μας. Όσον αφορά τη διαφάνεια για τα μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα, Χρειάζεται εδώ πέρα μια προσεκτική προσέγγιση και θεωρούμε ότι είναι προτιμότερη μια σταδιακή εισαγωγή υποχρεωτικών διατάξεων διαφάνεια για μια τόσο ευρύ ομάδα κατηγοριών στοιχείων ενεργετικού. Γι' αυτό τον λόγο θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τα, οι απαραίτητες δοκιμές ρευστότητας όσον αφορά το MIFID 2 και να μπορούν όλες οι μη μετοχικές κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού να υποφελούνται από ένα χαμηλότερο κατόφλι προσαρμοσμένο στο λόγο μέσο, όπου τα ζεύγια εντολών δεν θα απαιτούνται να έχουν προσυναλλακτική διαφάνεια. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε το απαιτούμενο επίπεδο προσυναλλακτικής διαφάνειας μόνο όταν τα χρηματοπιστικά αυτά μέσα είναι μικρότερου μεγέθους από ό,τι προβλέπεται στη σχετική πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να έχουμε λιγότερο αυστηρά κριτήρια για το πρώτο μόνο στάδιο. Έγινε μια πρώτη έρευνα όσον αφορά το πρότυπο αυτό και πρέπει να δούμε τι θα γίνει στα επόμενα στάδια του προτύπου. Αντίθετα με την πρόταση όμω αυτή, η ΕΣΜΑ θεωρεί στην γνωμοδότησή τη ότι πρέπει να περιλαμβάνονται εξ αρχή το πρότυπο και τα τέσσερα στάδια τη βαθμία αυτή εφαρμογή και να περιλαμβάνεται έτσι και η μετάβαση στο επόμενο στάδιο. Αν η ΕΣΜΑ τώρα εντοπίσει ότι υπάρχουν αντίξωε περιστάσει, τότε θα διακόψει τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο μέσω τροποποίηση του προτύπου. Πιστεύουμε ότι η προσέγγιση αυτή δίνει την καλύτερη δυνατή σαφήνεια και νομική ασφάλεια σε όλου του εμπλεκομένου και κατά αυτόν τον τρόπο λαμβάνουμε υπόψη και τη δικασία ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίση, κατά την άποψη τη ΕΣΜΑ, η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένω να μην ανταποκριθεί στη γενικότερη πρόθεση μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά ομολόγων ή μπορεί να το κάνει αυτό με μεγάλη καθυστέρηση. Οι απαιτήσει διαφάνεια στο πρώτο στάδιο βρίσκονται πολύ κοντά στι υφιστάμενε πρακτικέ. του να έχουμε τρει εδοχικέ διαδικασίε έγκριση μέσω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρό για όλου του εμπλεκομένου και ενδεχομένω να οδηγεί σε καθυστερήσει. Η πρόταση λοιπόν τη ΕΣΜΑ θα διασφαλίζει ότι τα συστήματα προφορική διαπραγμάτευση και τα συστήματα διαπραγμάτευση με πρόκληση υποβολή προσφορών θα μπορούν επίσης να υποφελούνται από τα νέα κατόφλια που προβλέπονται για τα μέσα αυτά και δεν θα έχουν όμως ανταγωνιστικό πλεονάκτημα σε σχέση με πλατφόρμες συναλλαγών οι οποίες θα μπορούσαν να ισχύουν επαόριστον. Όσον αφορά τώρα τα όρια θέσεων, επιβεβαίνουμε εδώ πέρα το αίτημα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο ευθυγραμμίζεται και με το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πρότυπο λοιπόν αυτό στην πράξη προβλέπεται ένα αυστηρότερο όριο του 2,5%, το οποίο μπορεί να εφαρμόζεται πλέον για τα γεωργικά παράγωγα, ενώ τα συμβόλαια περιορισμένη ρευστότητα μπορούν να αποφεληθούν από ένα υψηλότερο μέγιστο όριο. Η ΕΣΜΑ κατέληξε επίση σε κάποια μέτρα για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των δυνάμει αποκλεινουσών προσφορών παραδοτέων ομολόγων και να αντιμετωπιστεί επίση και το ζήτημα του αριθμού των ανοιχτών συμβολέων όταν περνάμε από το μη πλησιέστερο μήνα στον εγκύτερο μήνα παράδοση. Όσον αφορά τι προκλήσει μα, περιμένουμε στο μέλλον. Περιμένουμε ότι τα όρια περίπου 1.500 συμβολίων ρευστότητα θα πρέπει να θεσπιστούν από τι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ πριν από το 2018, όταν η ΕΣΜΑ θα πρέπει να υποβάλει και συγκεκριμένη γνωμοδότηση για κάθε τέτοιο συμβόλαιο για να εφαρμοστεί η MIFID 2. Έχουμε και το ζήτημα των παρεπόμενων δραστηριοτήτων. Η γνωμοδότηση της ΕΣΜΑ δεν διευθετεί το πολύ δύσκολο ζήτημα που έχουμε επιτάπητος, καθότι δεν προτείνουμε μια συγκεκριμένη δοκιμή βάση κεφαλαίων θεωρούμε ότι μια τέτοια δοκιμή, ένα τέτοιο τεστ παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Τα βασικότερα είναι ότι, τα, ότι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλόμενοι δεν παρέχουν τα κεφάλαια που προορίζονται για τη διαπραγμάτευση παραγόγων και επομένω σαν τέτοιο τεστ θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρό, ιδιαίτερα για του μικρότερου μη χρηματοοικονομικού παράγοντε. Επίση, τα κεφάλαια που χρειάζονται για τις συναλλαγές παραγόγων μέσω μη χρηματοοικονομικών αντισυμβαλωμένων αλλάζουν πάρα πολύ με την πάροδο του χρόνου. Επομένω, αν ακολουθήσουμε εδώ πέρα τι απαιτήσει τη ΜΥΦΙΤ, θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση ιδιαίτερα ασταθή. Παρ' όλα αυτά, προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μέθοδο μέτρηση προκειμένου να δημιουργηθούν τέτοια τεστ. Είπαμε ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω και να θέσουμε συγκεκριμένο κατόφλι, καθότι δεν έχουμε τα απαραίτητα δεδομένα για να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο κατόφλι. Επίση, είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε ένα ακόμα ζήτημα. Αν η θέσπιση δηλαδή ενό τέτοιου κατοφλίου είναι περισσότερο τεχνικό ζήτημα ή περισσότερο επιλογή πολιτική για το κατά πόσο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε δηλαδή τους μη χρηματοοικονομικού παράγοντες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Thank uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαγιόρ, επικεφαλή επικεφαλής ε, της μονάδας ε, για τις αγορές χρεογράφων. Καλημέρα σας και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας δίνετε αυτή η δυνατότητα να σας ενημερώσουμε για το πώς έχει η κατάσταση σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του ΜΥΦΙΤ 2. Ήδη έχουμε κάνει αρκετή δουλειά μετά από το σκρούτινι σλότ, οπότε και συναντηθήκαμε. Έχουμε εγκρίνει πλέον τον κατάλογο των κατεξοδότηση πράξεων, τρεις, δύο για το ΜΥΦΙΤ και μία για το ΜΥΦΙΤ και είναι τώρα στη φάση του ελέγχου από το Κοινοβούλιο και βέβαια με τα χαράς να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που ενδεχομένως έχετε σε σχέση με ορισμένε από τις επιλογές πολιτικής που περιλαμβάνονται σε αυτές τις κατεξιοδότηση πράξεις. Για να είμαστε και μετεροπαθείς, κοντεύουμε να φτάσουμε στο αμισά του δρόμου σε ό,τι αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα. 16 έχουμε ήδη εγκρίνει και θα εγκρίνουμε τα περισσότερα, αν πάνε όλα καλά και βάσει με το πρόγραμμα, πριν από τις θερινές διακοπές. Ίσως να έχουμε κάποια μικρή καθυστέρηση σε ένα από τα τρία γιατί χρειάστηκε ένας δεύτερος γύρος. Και βέβαια εδώ έρχομαι στον πυρήνα των πολιτικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί τα τρία RTS. Ανέφερε ήδη τα σχετικά ο πρόεδρος της ΕΣΜΑ. Δεν θέλω να επισέλθω στις τεχνικές λεπτομέρειες. Με τρεις προτάσεις μόνο θα σας εξηγήσω ποια είναι η συλλογιστική του σώματος των επιτρόπων πίσω από την απόφαση τα τρία αυτά πρότυπα να γίνουν αντικείμενο ενό δεύτερου γύρου. Οι επίτροποι έκαναν ένα βήμα πίσω και εξέτασαν τη συνολική εικόνα. Δηλαδή, πώς έχει η ευρωπαϊκή οικονομία, τι πρέπει να γίνει για να έχουμε μεταρρυθμίσεις που θα έχουν νόημα, που θα μπορούσαμε να επιφέρουμε σωστές διορθώσεις, αλλά να μην χαλάσουμε και αυτά που δουλεύουν μέχρι στιγμής σωστά. Φυσιολογικά η εστίαση αν έχουμε μια πιο γενική οικονομική προσέγγιση, είναι στα εταιρικά ομόλογα, τα οποία είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, ε, ε, για να μπορέσουν να συλλέξουν κεφάλαιο οι εταιρείε. Άρα πρέπει να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε μια εύρυθμη αγορά σε αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό και θέλουμε ένα χρονοδιάγραμμα σταδιακής ένταξης, phasing schedule. Συνεργαζόμαστε στενά με την ΕΣΜΕ για να βρούμε τα σωστά benchmarks για αυτά τα ε, benchmark, για αυτά τα ομόλογα, ώστε να έχουμε διαφάνεια. Θα πρέπει να δούμε πόσα ε, ομόλογα πειράζονται από διαφάνεια και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Θεωρούμε δυνάμει, μάλλον υπό το πρίσμα των οικονομικών συνθήκων και της μακροοικονομικής ε, κατάστασης, θέλουμε να έχουμε μία ολιστική προσέγγιση και μετά να περάσουμε το ένα στάδιο στο άλλο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι χρηματοδοτικέ τάσει, να αξιολογήσουμε την ρευστότητα τη αγορά και να εθετήσουμε μια ε, σόφρονα απόφαση όταν θα χρειαστεί να περάσουμε το ένα στάδιο στο άλλο. Και ο πιο λογικό τρόπο για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα είναι πρώτα να έχουμε την έκθεση και μετά την απόφαση για μετάβαση στο άλλο στάδιο. Και έπειτα θα εγκριθεί το νέο και θα υποβληθεί στο δημοκρατικό έλεγχο ε, από το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τα παράγωγα ε, στις σίγουρα έχουμε κάποια τρόφιμα και πρώτες πολύ ευαίσθητες. Χαιρετίζουμε την εισαγωγή ενός κατώτερου κατοφλίου για κάποιες συμβάσεις που αφορούν για αγροδιατροφικά προϊόντα. Επίσης, ό,τι αφορά τις, ε, τα πρότυπα για τις παρεπόμενες δραστηριότητες, θέλουμε να πετύχουμε. Είναι μεγάλη πρόκληση. Πρέπει να δούμε στο μέλλον πόσες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες θα υπόκεινται στην εξουσιοδότηση MIFID και αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις ε, που ξεπερνούν τις κεφαλαϊκές απαιτήσει εταιρείε MIFID. Θέλουμε και εδώ λοιπόν να βρούμε τη σωστή λύση. Καλωσορίζουμε τη γνωμοδότηση της ΕΣΜΑ δεν είναι σχέδιο RTS, άρα πρέπει να κάνουμε και εμείς τώρα πολλή δουλειά και θα την κάνουμε. Έχουμε την ε, τεχνογνωσία και την εμπειρία, έχουμε ε, τις γνώσεις, μπορούμε να αξιολογήσουμε τις διαφορετικές επιλογές που μας ε, υπέβαλε ως πρόταση η ΕΣΜΑ. Πέντε τον αριθμό επιλογές έχουμε στη διάθεσή μας για τη δοκιμή των παρεπόμενων δραστηριότητων. Πέντε επιλογές για τον ορισμό του τι είναι ε, trading activity, speculative trading activity και δύο για το είναι, τι είναι basic trading activity. Και θα πρέπει με βάση όλα αυτά να ορίσουμε ένα λόγο, ένα ratio. Θα μελετήσουμε πολύ προσεκτικά τις διαφορετικές επιλογές, για να δούμε τι είναι speculative trading activity και μετά θα δούμε και θα ζυγίσουμε τις διάφορες επιλογές για να δοθεί το κεφάλαιο στις βασικές δραστηριότητες. Τώρα, Πιστεύουμε ότι πρέπει να διαδραματίσει ένα ρόλο και κατανοούμε το κεφαλαίο μεταξύ των δύο δραστηριοτήτων στο επίπεδο 1. Επίση, το κεφάλαιο δεν είναι η μόνη δοκιμή, δεν είναι το μόνο τεστ, γι' αυτό και έχουμε και μια γενική ε, δοκιμή για τα μερίδια τη αγορά. Θέλουμε το σύντομα το δυνατόν να επεξεργαστούμε αυτό το πρότυπο και αν υπάρξει καθυστέρηση, θα υπάρξει μάλλον μόνο για αυτό το πρότυπο, επειδή χρειάζεται να γίνει ουσιαστική δουλειά ακόμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λούτερς. Ο εισηγητής έχει το λόγο και θα μιλήσω γερμανικά πραγματικά τώρα. Sorry for that. Πρώτα απ' όλα λοιπόν σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση των όσων είχαμε μέχρι στιγμής υποβάλει. Θεωρώ πως είχαμε ένα μύθιτ το οποίο ήταν κάπως ε, γρήγορο, μια γρήγορη λύση και τώρα στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις ε, αγορές και εδώ πέρα θέλω να ευχαριστήσω του ε, συναδέλφου. Δεν πίστευα ότι θα τα καταφέρναμε τόσο γρήγορα. Ήμασταν στον τριμερή διάλογο γρηγορότεροι ε, από τις ε, προτάσεις των άλλων συνομοθετών. Αλλά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, είχαμε υποσχεθεί, μας είχαν υποσχεθεί ότι θα ήταν όλα έτοιμα μέχρι την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Κάποια πράγματα λοιπόν θα ήθελα να αναφέρω όσον αφορά την παροχή ε, συμβουλών. Είχαμε αναφέρει έναν κατάλογο με παραδείγματα που βελτίωναν την ποιότητα και μία πρόταση ήταν να αναφερθούν ρητός ε, ορισμένες περιπτώσεις, κάτι το οποίο δεν συνέβη και δεν ξέρουμε γιατί η Κομισιόν δεν θέλησε να επεκτείνει την λίστα. Όσον αφορά επίσης το άρθρο 76 αναφέρεται ξεκάθαρα πως οι τελο... τηλεφωνικές ε, καταγραφές και καταγραφές ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν ε, την πολυπλοκότητα των συναλλαγών αυτών. Επίσης θα πρέπει να καλύπτουν και τα σημαντικά εσωτερικά τηλεφωνήματα και εσωτερική ηλεκτρονική επικοινωνία. Εγώ θεωρώ πως θα πρέπει και τα τηλεφωνήματα και τα πρακτικά ε, διαφόρων τέτοιων συνεδριάσεων ε, να θεωρηθούν εξίσου σημαντικά, κάτι το οποίο δεν ίσχυε για την εσωτερική επικοινωνία, αλλά θα πρέπει η Κομισιόν να δεχτεί την σημαντικότητα των ε, δύο αυτών περιπτώσεων όπως περιγράφεται στο επίπεδο 1. Επίσης, για εμάς είναι σημαντική η διευκρίνηση και η ερμηνεία από τις εθνικές εποπτικές αρχές, όπως αναφέρεται εδώ πέρα ε, το τι γίνεται με τις Commission Sharing Agreements έχουμε αναφερθεί σε δύο μεγάλα κράτη-μέλη που κατέληξαν σε τελείως διαφορετικές ε, ερμηνείες ότι μια πρακτική είναι και δεν είναι ε, ταυτόχρονα δυνατή. Επίσης, ε, ανάλυση της αγοράς ε, στόχου. Στην MIFID 2 νομίζω πως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα ή αυτό είναι κάτι το οποίο καθαρίζει, καθορίζει ο παραγωγός και όχι αυτός ο οποίος πωλεί το προϊόν. Στο άρθρο 10 αναφέρεται πως οι εταιρείε καθορίζουν την αγορά στόχο ακόμα και αν δεν έχει καθοριστεί αγορά στόχος από αυτόν ο οποίος επινόησε το προϊόν. Ποιος είναι τελικά ο υπεύθυνο μετά. Έχουμε το θέμα του καθεστώτος για την συστηματική υιοθέτηση για να δούμε ποια θα είναι τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο επίπεδο 1 έχουμε καθορίσει ως ε, κριτήριο το ότι θα πρέπει να υπάρχει συστηματική και συχνή χρήση. Και θα πρέπει να μην υπάρχει συχνή αλλαγή του καθιστώτος κατόπιν. Το Κοινοβούλιο πρότεινε για μέσα τα οποία δεν αφορούν το ίδιο το ίδιο κεφάλαιο να εισαχθεί μια ρύθμιση de minimis, ειδικά για τους ε, μικρότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ε, δεν ακολούθησε αυτή την πρόταση Κομισιόν και θα ήθελα να μάθω γιατί ένα άλλο θέμα το οποίο βλέπω επικριτικά είναι η ρήτρα One Triggers All για συστηματική εσωτερικοποίηση του κινδύνου. αν ε, πληρούνται τα κριτήρια παραδείγματο χάρη για δανεισμό, θα πρέπει να ισχύει αυτό για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα τη ιδία ε, τάξη. Εδώ πέρα έχω σοβαρέ αμφιβολίε για το εάν η προσέγγιση αυτή συμφωνεί με τον ορισμό του άρθρου 421 της ε, MIFID που μιλάει μόνο για συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα. Επιπλέον τίθεται το ζήτημα του πώς καθορίζονται οι διάφορες τάξεις χρηματοπιστωτικών μέσων. Επιπλέον το Κοινοβούλιο ζήτησε διευκρινήσεις ε, για το ότι δεν επιτρέπεται match principal trading για SIs όπου ισχύει το άρθρο 4 38 της ε, MIFID 2 η Κομισιόν δεν δέχτηκε αυτόν τον ορισμό στο εκτιμώντας 19 και προτίμησε να πάει σε ένα εσωτερικό σύστημα σε πολυμερή βάση. Γιατί η Κομισιόν δεν δέχτηκε την σαφή διατύπωση του επίπεδου 1 μετά position limits, ε, διαφάνεια και μέσα τα οποία δεν είναι ιδίου κεφαλαίου και εδώ πέρα κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, η Κομισιόν απέστειλε τρεις προτάσεις ρυθμιστικών στάνταρτ ξανά πίσω στην ε, ΕΣΜΑ. Θα περιοριστώ σε λίγα από αυτά. Η γνωμοδότηση της ΕΣΜΑ θεωρώ πως είναι ιδιαίτερως προβληματική. Αφενός η ΕΣΜΑ σε αντίθεση με τα όσα επιθυμούσαμε εμείς ε, και η Κομισιόν νομίζω δεν ζήτησε να υπάρξει ένα τεστ το οποίο θα βασίζεται στο κεφάλαιο το οποίο μετά όμως ε, προσπαθεί και μας λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει χωρίς να κάνει κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Τι σημαίνει αυτό, τι θα κάνει η Κομισιόν με την ε, πρόταση αυτή. Πραγματικά προσπάθησα να περιοριστώ στα σημαντικότερα μόνο και με συγχωρείτε αν μακρηγόρησα. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα ακόμα και ελπίζω να λάβουμε κάποιες απαντήσεις σήμερα. Σας ευχαριστώ. Next Επόμενος ομιλητής για τους σοσιαλδημοκράτες είναι ο Πολ Τάγκ. Σωστά, ναι. Ευχαριστώ. Να μιλήσω εκ μέρους της αναλύς Dodge. Είναι στην εκστρατεία και ελπίζουμε να είναι επιτυχής. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους και οδησηγητές. Συνεργαστήκαν πολύ καλά. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Νέα εργάστηκαν σκληρά για 30 περίπου νομοθετήματα επίπεδου 2. Ποιο είναι το γενικό πλαίσιο. Τρία βασικά θέματα θέλω να αναφέρω. Πρώτο, τα όρια θέσεως για τα παράγωγα. Εμείς εκφράσαμε ανησυχία για την αρχική πρόταση της ΕΣΜΑ. Χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει τις τεχνικές προδιαγραφές. Κάποιες από τις αναθεωρήσεις ΕΣΜΑ είναι ευκρόστιχες, οπότε τα κατώτερα όρια να φτάσει στο 2,5% για τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα. Κάποια άλλα στοιχεία όμω είναι λιγότερο πρόσδεκτα. Η απόφαση, το ανώτατο όριο του καθεστώτος να πάει στο 50% για κάποια συμβάση σημαίνει ότι ένα φορέ στην αγορά μπορεί να ελέγχει ε, το μισό ποσό αυτών των προϊόντων. Απαράδεκτο και δεν τηρεί και την πολιτική συμφωνία του επίπεδου 1. Ταυτόχρονα, η ΕΣΜΑ κράτησε τα βασικό όριο στο 25%. Εμεί σοσιαλιστέ πάντα λέγαμε ότι πιστεύουμε σε αυτόν τον αριθμό. Ότι έπρεπε να είναι μικρότερο το ποσοστό. Η βάση θα πρέπει να στέλνει μήνυμα στου εθνικού ρυθμιστικού φορεί. Τα, τα όρια πρέπει να είναι στο χαμηλότερο επίπεδο για τα βασικά προϊόντα για να σταματήσουμε την κερδοσκοπία και τη στρέβωση των προϊόντων όπως είναι τα κάψιμα και τα προεκπαιδευτικά. Η ΕΣΜΑ δεν συμπερίλαβε για τις διάφορες κοινοφιλείς υπηρεσίες ε, όρια θέσεων. Αυτό εμπεριέχει το στοχικό έγγραφο συζητήσεων, αλλά διαγράφει. Τέτοια διαγραφή παραβιάζει το επίπεδο 1. Εκεί αναφέρεται ότι για τι κοινοφελεί υπηρεσίε οι ρυθμιστικέ αρχέ πρέπει να λάβουν υπόψη τα όρια. Πάμε τώρα σε αυτά που θέλουμε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά που τονίσαμε να εξετάσει. Πριν επιστρέψουν οι προδιαγραφές σε εμάς τελικά για έγκριση ή απόρριψη. Δεύτερον, παράγωγα των βασικών αυτών προϊόντων. Είναι οι δοκιμές των βοηθητικών δραστηριοτήτων. Ο τελικός κανονισμός πρέπει να εξασφαλίσει ότιμου όρου μεταξύ μοτοστικών εταιριών που κερδοσκοπούν στην αγορά παραγόγων και των εταιριών πρώτων υλών, αν θέλετε, των βασικών προϊόντων που έχουν τόσο μεγάλα κέρδη που ουσιαστικά είναι επενδυτικοί φορεί. Τα όρια της δοκιμέ θα πρέπει να τόσο ψηλά μάλλον είναι πολύ ψηλά και μπορούν να εξαιρούνται κάποιες εταιρείε. Πρόθεση του MIFID 2 ε, όμως ήταν να καλύπτονται. Τρίτον, επενδυτικές έρευνες. Καλή προσπάθεια Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έσμα για συμβιβασμό. Να υπάρχει αποδέσμευση του κόστους. Να έχουμε πιο διαφανές καθεστώς. Ακούσαμε όμως φήμες ο τελικό άρθρος, το άρθρο θα ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως από διάφορους ρυθμιστικούς φορείς όσον αφορά την εφαρμογή αυτού. Οι ρυθμιστικοί φορείς κρατών μελών φρονούν ότι όλες οι διευθετήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να τροποποιηθούν για να συμμορφωθούν με το νέο καθεστώς. Άλλοι ρυθμιστικοί φορείς λένε στους συμμετέχοντες στην αγορά ότι λέει κανόνες επιτρέπουν τη συνέχιση της καθεστικίας τάξης. Αυτό είναι απαράδεκτο θα είναι επιβλαβέ όσον αφορά τι σηματοστατικές εταιρείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει προσανατολισμού στου ρυθμιστικού φορεί, αναφέροντα ρητά το τι γίνεται με τι ευθετήσεις όσον αφορά ε, ε, τα διάφορα μερίσματα που θα παίρνουν οι εταιρείε. Είναι ο μόνο τρόπο να εξασφαλίζουμε κάποια συνέπεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα βοήθησε, την ευχαριστούμε, αλλά περιμένουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις που έχουν σε αυτά τα τρία σημεία που έθεσα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πολ. Και τώρα και η Swinburne έχει το λόγο για το ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ομάδα της ΕΣΜΑ. Εργάζονται σκληρά για το MIFID και το MIFIR. Εκτιμούμε τη σκληρή δουλειά που έγινε. Αλλά έπρεπε να βρούμε και σωστή λύση. Γι' αυτό χρειαζόταν συνεργασία που την εκτιμώ. Ευπρόσδεκτη διαβεβαίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα επιλέξει να μην υπάρχει αυτοματισμός όσον αφορά το καθεστώς διαφάνειας για τα εισοδήματα προ-συναλλαγών. Καλωσορίζουμε λοιπόν την πρόταση της ΕΣΜΑ για την ετήσια αυτόματη αύξηση. Το επιβεβαιώνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως παρανόησα αυτόματες αυξήσεις, κατά την άποψή μου, την αξιολόγηση ευστότητας θα την καθιστούν άχρηστη. Διότι θα υπολογίζεται το αποτέλεσμα πριν γίνει η προσπάθεια. Και το Κοινοβούλιο δεν θα μπορεί να ελέγχει αυξήσεις στις υποχρεώσεις περί διαφανείας. Περί αυτού πρόκειται, αυτό θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά το να μην υπάρχει αυτοματισμό στον υπολογισμό. Όμως, ακούγοντας τα λεπτομερή σχόλια της ΕΣΜΑ για τα όρια θέσεων και τα διάφορα σχόλια Έχω διαφορετική θέση. Καλωσορίζω την προσέγγιση της ΕΣΜΑ. Κυρίως το μηχανισμό για τους μήνες σποτ με μη σποτ. Έκαναν ένα δύσκολο συμβιβασμό να λειτουργεί στα πλαίσια της λύσης. Όσον αφορά αυτά τα όρια των θέσεων είμαι πιο ικανοποιημένη τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Με ικανοποιεί η προσέγγιση της σχόλια σε άλλο τομέα. Στο μέλλον, τα παρα... παράπλευρα προϊόντα, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Μας προσέγγισαν διάφορες φορείς να βρούμε λύση. Έχει προβληθεί το θέμα και στον τύπο. Τα θέματα που θίγονται σε επιστολές και στον τύπο ότι πολλοί θεωρούν ότι δεν έχουν εισακουστεί και δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για το μύφη δεν λησμονούν τους τριμερείς διαλόγους. Το συζητήσαμε εκτενώς το θέμα. Και δεν υπήρχε ζήτηση για ενοποιημένο αρχείο. Και δεν θα έπρεπε να ανησυχούμε. Εγώ έχασα όσον αφορά την τοποθέτησή μου, έπρεπε να συμβιβαστούμε. Δεν έχουμε εγγυηθεί ένα ενοποιημένο πλαίσιο στο επίπεδο 1 και δεν έχουμε βάλει ελέγχου τιμών όσον αφορά τα στοιχεία. Τα περισσότερα θέματα που θίγονται όσον αφορά τα στοιχεία δεν μπορούν να καθορίζονται στο επίπεδο 2. Διότι τα συζητήσαμε στο επίπεδο 1 και δεν τα προσεγγίσαμε όπως απαιτεί Άρα θα πρέπει αυτή με τα, οι φορεί των παραπλεύρων αυτών προϊόντων να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσει. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΣΜΑ θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν για να εισακουστεί η φωνή των επενδυτών σε όλες τις φάσεις για τη διαμόρφωση προτάσεων. Τέλος, κάτι που έθιξε ο Πολ Ταν. Πώς ξεκαθαρίζουμε τις ερμηνείες όσον αφορά την ενή αγορά για τα RTS Σαν διαπραγματευτική ομάδα θέσαμε εκτενή ερωτήματα. Μήπως έπρεπε να δημοσιοποιηθούν κάποιες απαντήσεις, ούτω ώστε να καθησυχάσουν και οι έξω. Και αν δεν αρκεί αυτό, ίσως με κάποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΣΜΑ επισήμως να εκδώσουν ερωταπαντήσεις για να διευκρινίσουν κάποια θέματα. Δεν θα πρέπει ένας τομέας να απαγορεύει την έρευνα, τις συμβάσεις για έρευνα και άλλος τομέας να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Τέλος, κάτι που ήταν μεγάλο βήμα για το Κοινοβούλιο. Συζητήσαμε τις απαιτήσει περί πληροφοριών στο MIFID. Θα θέλαμε να υπάρχουν έγγραφα όσον αφορά τα, ε, τις διαπραγματεύσεις του ε, επίπεδου 1. Αντί για χαρτί είπαμε ε, να εγγράφονται τα στοιχεία σε κάποιο μέσο διαρκείας. Κινούμεθα από ψηφιακή αγορά και θέλουμε ψηφιακή ενιαία αγορά. Άρα έπρεπε να καταλάβουμε ότι κάποτε στο μέλλον δεν θα χρησιμοποιείται πια το χαρτί τόσο εκτενώς. Εκπλαγήκαμε λοιπόν που είδαμε ότι από τα μέσα διαρκείας, τα ανθεκτικά μέσα πήγαμε στο χαρτί ξανά σε αυτή την αναφορά στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφού αλλάξαμε και πήγαμε από έγγραφα σε ανθεκτικά μέσα, μήπως να το διορθώσουμε ξανά αυτό. Όταν θα έχουμε ψηφιακές πηγές πληροφοριών και τα πάντα ψηφιακά, να μην πρέπει να επανέλθουμε ξανά στη χρήση του χαρτιού. Ευχαριστώ πολύ και η, φιλελεύθερη. Κόρα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΣΜΑ. Έκαναν πολλή δουλειά. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους κοιόδης. Εστιαζόμενοι επί των προβλημάτων που απομένουν, λησμονούμε την καλή δουλειά που έγινε. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Τεράστια προσπάθεια έγινε. Όμως, δυστυχώς δεν είναι τα πάντα επιτάπητος όπως αναμενόταν. Ο συνήθως, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες αφορούν τα όρια και τους ορισμούς. Και εκεί δημιουργούνται μεγαλύτερα προβλήματα. Δεν θέλω να επαναλάβω τα καλυφθέντα ζητήματα και τις ερωτήσεις που έθεσαν ο εισηγητής και οι σκιώδης για τη σαφήνεια που λείπει ακόμα όσον αφορά τις δυνατότητες ερμηνείας διαφόρων διατάξεων. Θα ήθελα να προσθέσω μια ερώτηση. Και εγώ έχω την ίδια απογοήτευση όπως και καίει. Κάποια συμπεφωνηθέντα στο επίπεδο 1 δεν μπορούν να καθοριστούν στο επίπεδο 2. Εγώ δεν ήμουν παρούσα στα συζήτηση του επίπεδου 1 και δεν μπορώ να επηρεάσω πλέον αυτά που φασίστηκαν. Έχουμε ακόμα προβλήματα ανεπίλητα και δεν θα ήθελα να κινηθούμε σε επίπεδο ανώτερο, όπως το επίπεδο 3, όσον αφορά τα CSAs. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Αναφερόμενοι στα προβλήματα, με τις διάφορες προδιαγραφές για τις επικουρικές δραστηριότητε. Είναι σημαντικό αυτό σαν θέμα. Πρέπει να το λύσουμε. προχωράτε συνετά. Το καταλαβαίνω, είναι πολύ σημαντικό. Όμως, να τονίσω ότι πρέπει να λύσουμε τις εκκρεμότητες στο επίπεδο 2. Αυτά είχα να πω πάνω κάτω για την ώρα και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κόρα. Δεν βλέπω κάποιον της Γκουέ να παρίσταται. Σβέν Γκίγκολτ από τους Πράσινους συνεχίσω αγγλικά. Ευχαριστώ εκ νέου. Ευχαριστώ την ΕΣΜΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τους ευχαριστώ για τη δουλειά τους και για τη συζητήση μεταξύ θεσμικών οργάνων. Και διότι έλαβαν υπόψη κάποια από τα θέματα που θίξαμε. Να πω καταρχάς το εξής. Βλέποντας προστασία επενδυτών και καταναλωτών, αποδυναμώθηκε κάπως το αρχικό κείμενο της ΕΣΜΑ και με την πάροδο του χρόνου εντός των διαδικασιών της ΕΣΜΑ υπήρξε κάποια αποδυνάμωση και δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτό και να αυξηθεί στα τελικά στάδια. Θα επικεντρωθώ επί των ορίων θέσεων παρόλο που εύχομαι καλή τύχη στην ΚΕΙ αυτές τις ημέρες Πρέπει να πω ότι αν λέει ο Σαφάτσε Ορίων ότι είναι πιο ικανοποιημένη τώρα από ό,τι ήταν κατά το παρελθόν, αυτό με κάνει να ανησυχώ. Αρχές Μαΐου ε, εξέδωσε γνωμοδότηση ΕΣΜΑ με τις προδιαγραφές ε, για τα όρια θέσεων RTS 21. Αν συγκρίνουμε αυτό με αυτά που ζήτησε το Κοινοβούλιο, τι βλέπουμε παραμένει σημαντικό πρόβλημα για να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε ως νομοθέτες. Το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε στην επιστολή του και παραθέτω το καθεστώς να στέλνει σαφές μήνυμα προς εθνικές αρμόδιες αρχές ότι θα πρέπει να καθορίσουν κατώτατα όρια θέσεων όποτε το επιτρέπει η ρευστότητα. Και αυτό δεν ισχύει. Η ΕΣΜΑ τροποποίησε το κατώτατο όριο από 5% σε 2,5% αλλά αφήνει την βασική γραμμή, τη βάση, όπως είπε και ο Μπόλταν, στο 25 σαν βάση και 35% ανώτατο όριο και τα άφησα μετάβλητα. Το κατώτατο όριο δεν θα ισχύει μόνο για περιορισμένο αριθμό προϊόντων, ε, παραγόγων βασικών προϊόντων όσα είναι συμβάσεις πάνω από 50.000 παρτίδες ε, για παραπάνω από μια τρίμηνη περίοδο καλύπτονται από αυτό. Αυτές οι συμβάσεις πρέπει άμεσα να συνδέονται με ανθρώπινη κατανάλωση. Άρα θα πρέπει να θεωρούνται τα προϊόντα αυτά σαν τρόφιμα προς ανθρώπινη κατανάλωση. Άρα βασικά προϊόντα και οι τιμές των τροφίμων συνδέονται πολύ στενά, όπως είναι οι ζωοτροφές και η ενέργεια όμως εξαιρούνται προειδοποιώ ότι δεν πρέπει να ακολουθήσω αυτή την προσέγγιση. Για να το πω, μα, αν οι αγορέ κάποια στιγμή είναι πολύ ρευστέ, μπορεί να σκοτώσει ανθρώπους όχι μόνο από στέρηση από τα τρόφιμα, αλλά και επηρεάζοντα ε, την ενέργεια και τις ε, ζωοτροφές που χορηγούνται στα ζώα. Δεύτερον, το Ευρωκοινοβούλιο πρότεινε να Έχουμε την παροχή των προϊόντων για, για μηνιαία όρια μη σποτ. Και είχαμε ζητήσει να καθοριστούν αρχ... τα όρια αρκετά χαμηλά. Η ΕΣΜΑ συμπεράβε στο νέο σχέδιο κειμένου ένα RTS και σύσταση στους αρχές να προσαρμόσουν προς τα κάτω τις θέσεις ορίων προς τα κάτω ή προς τα άνω αν το συμφέρον είναι, το ενδιαφέρον είναι ανώτερο ή κατώτερο από ότι αυτά που παραδίδονται και καθορίζονται όρια διευρύνοντας τον ορισμό των αυτοπαραδομένων προϊόντων. Υποκατάστατα προϊόντα, πρώτε ύλες επίση συμπεριλαμβάνονται. Είχαμε ζητήσει μετά οι συμβάσεις που συνδέονται στενά με οικονομικά αποτελέσματα θα πρέπει να καθορίζονται από τα ίδια όρια θέσεις Αλλάζει του ορισμού η ΕΣΜΑ όσον αφορά τι οικονομικά αντίστοιχε συμβάσει οτιέ, που σημαίνει ταυτόσημα εκτό από διαφορετικέ προδιαγραφέ για το μέγεθο παρτίδων και ημερομηνίε παράδοση που ε, παρεκκλίνουν περισσότερο από μία ημερολογιακή ημέρα. Αυτές είναι ελάχιστε οι αλλαγέ και δεν μπορούν να επηρεάσουν το να μην τηρούνται τα ωριά μας. Τέλος, το Κοινοβούλιο επανειλημμένα είπε ότι η πτητικότητα είναι παράμετρος που θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις προδιαγραφές σύμφωνα με την εντολή του επίπεδου 1. Η ΕΣΜΑ για μια ακόμη φορά αγνόησε τη ρητή νομοθετική εντολή που της ανατέθηκε και δεν μπόρεσε στην πτητικότητα των αγορών τη δυτικότητα των αγορών να τη λάβει υπόψη στη μεθοδολογία που προτείνει. Βάσει όλων αυτών και έχοντας υπόψη ότι η παράγραφος 7 του άρθρου 57 του ΜΥΦΙΔ σαφώς απαιτεί ότι πρέπει να υπάρχει ομοιόμορφη και κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των ορίων θέσεων, ότι όλα αυτά υπολείπονται των αναμενωμένων από πολλούς πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της μεγάλης, των μεγάλων αλλαγών όσον αφορά τα κρίσιμα βασικά προϊόντα που είναι αρκετά ρευστά σαν αγορές για να ρυθμιστούν. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα και να συμπεριλάβει στις προδιαγραφές σαφείς προτάσεις για τις προβλεπόμενους ετησίους ελέγχους της εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο από τις αρμόδιες αρχές και πώς θα στεδιαστεί αυτό το κατάλληλο πλαίσιο. Κάτι που δεν διευκρινίζεται ακόμα στα RTS. Ευχαριστώ πολύ Σβέν. Πολλές ερωτήσεις ετέθησαν πολλά θέματα, περιμένουμε απαντήσεις. Ο Στίβεν Μαϊόρ έχει το λόγο από την ΕΣΜΑ. Ευχαριστώ Μάρκους. Θα είναι δύσκολο, λαμβανωμένο υπόψη του χρόνου, να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω όμως και θα ζητήσω από τον Τρίκο Μπιονοβεντούρα να απαντήσει στο θέμα των ορίων θέσεων. Μία-δύο γενικές απαντήσεις να δώσω. Ευχαριστώ πολύ όσους έκαναν σχόλια και όσοι υπέβαλαν ερωτήσει σχετικά με το έργο. Θα εστιαστώ των RTS, γιατί νομίζω ότι οι κατεξιδότητες συμπράξει αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να απαντήσω ότι ε, ξεκινάμε την επεξεργασία των προσανατολισμών του επίπεδου 3. Δηλαδή, μετά θα έχουμε κάποιες νομοτήσεις αργότερα για να υπάρχει συνέπεια στην εφαρμογή των επιπέδων 1 και 2. Αυτό εφήγει στα πλαίσια τη Συμφωνία Επιμερισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Σχετικών Διευθετήσεων. Και το θέμα είναι σε ποιο βαθμό τα επιτάπη το συνάδουν με αυτό. Θα πρέπει καταρχά να αναγνωρίσουμε το εξή: Ότι τη στιγμή θα ξεκινήσει το MIFID πρέπει να υπάρχει συνέπεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τακτικά μέτρα του επίπεδου 3 για να εξασφαλίζουμε συνέπεια. Απαντώντα την ερώτηση αν αυτό συνάδει με το CSA ή όχι, αυτό είναι δύσκολο, δεν μπορεί να απαντηθεί διότι το CSA δεν καθορίζεται νομικώς σαφώς. Αυτό που θεωρούν κάποιοι ότι είναι CSA ίσως να ποικίλει από χώρα σε χώρα. Ποιο είναι ο αποφασιστικό παράγοντα, Είναι αυτό που περιέχεται στα επίπεδα 1 και 2. Και ότι το CSA αυτό καθε αυτό δεν καθορίζεται, δυσχεραίνει κατά πολύ την απάντηση. Άρα χρειάζεται αξιολόγηση κατά περίπτωση. Ε, νομίζω ότι όσον αφορά αυτά που υπόθηκαν για την συμμετοχή των φορέων των παραπριόντων σε επίπεδο ΕΣΜΑ συμμετέχουν στις προσπάθειές μας, συμμετέχουν στην ομάδα των ενδιαφερομένων, συμμετέχουν στις βουλευτικές ομάδες ε, και γενικά βρίσκουν το δρόμο τους όταν θέλουν να σχολιάσουν αυτό που κάνουμε. Τα άλλα θέματα που αναφέρθηκαν, στα οποία θέλω να απαντήσω. Καταρχάς, για τη διαφάνεια για τα, τις βοηθητικές δραστηριότητες μάλλον πρώτα απ' όλα. Να πούμε ότι το επίπεδο 1 προέβλεπε ότι η δοκιμή βάση κεφαλαίου ήταν δυνητικά ε, εφαρμόσιμο. Δεν ήταν ρητό το προπετούμενο. Ξεκινήσαμε λοιπόν στις διαβουλεύσεις, στις πρώτες διαβουλεύσεις ε, με τις δοκιμές ε, βάση κεφαλαίου αλλά θεωρήσαμε ότι υπήρχαν αδυναμίες όσον αφορά τις δοκιμές, σχετιζόταν με τη διαχείρισή του, ε, οπότε ήταν δύσκολο να το χειριστεί κανείς και είναι μέθοδος ασταθής, δηλαδή ποιο κεφάλαιο συμμετέχει στο εμπόριο παραγόγων και αυτό μας έλεγαν εξάλλου και οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι κύκλοι στις διαβουλεύσεις. Δηλαδή ότι διέβλεπαν προβλήματα. Γι' αυτό δεν βαστήκαμε στο κεφάλι στις δοκιμές, όμως υπάρχει πολιτική απέτηση για κάτι τέτοιο και γι' αυτό ε, ξεκινήσαμε αυτές τις δοκιμές, δώσαμε κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν είχαμε πολύ χρόνο και έτσι δεν ολοκληρώσαμε την προσέγγιση και τις δοκιμές. Και δεν βρήκαμε πλήρη λύση. Τέλος, τη διαφάνεια όσον αφορά τα... τις άλλες διεργασίες που δεν αφορούν τα αξιογράφα. Θέλαμε επόμενες, ε, τα επόμενα στάδια να συμπεριφθούν στις προδιαγραφές. Θέλουμε να δούμε τεχνικώς τι γίνεται με τη ρευστότητα των αγορών. Έχουμε και εργαλεία και δυνατότητα σαν έσμα να κάνουμε αξιολόγηση ρευστότητα των αγορών. Πιστεύουμε ότι αν αυτό γίνει σωστά, μπορείς να σταματήσεις τη διαδικασία. Και αν κινηθείς γρήγορα, συνεργασία ΕΣΜΑ, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και θεσμικών οργάνων, αν υπάρχει συνεργασία, αποφεύγουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση αν δούμε ότι η αξιολόγηση ρευστότητα ε, προβλέπει ε, προβλήματα για τις αγορές. Θα σταματήσω εδώ και να δώσω το λόγο στο Ροντρίγο Μπουενοβεντούρα για το επόμενο θέμα. Σύντομα, γιατί δεν θα μπορέσω να αναφέρω λόγω του πετρεσμένου χρόνου τα πάντα. Θα ήθελα να εστιάσω στο θέμα των διακυμάνσεων ε, της ρευστότητας ε, ασάφειας. Ε, πράγματι, έχει θεωρηθεί ως ένας παράγον αρχικά που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη, τουλάχιστον στην πρώτη διαβούλευση για τα όρια Αναλύσαμε όμως ε, κάποια στοιχεία και με τις απαντήσεις που λάβαμε και στις διαβλέψεις δεν βρήκαμε να υπάρξει στατιστική σχέση μεταξύ αυτής ε, της διακύμανσης ε, και καταχρηστικής ε, ε ισχύω της αγοράς. επομένως θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για τα υψηλότερα ή χαμηλότερα όρια αυτό το κριτήριο. Στα γεωργικά προϊόντα, για παράδειγμα, υπήρξαν λίγο, υπήρξε μικρότερη ρευστότητα στη μέσα ε, ιδίω κάποια τρίμα του προηγούμενου έτου. Και αν είχαμε συμπεριλάβει υψηλότερη, υψηλή ρευστότητα ή ασάφεια διακυμάνσεις ε, ίσως χαμηλότερα όρια, εκεί θα είχαμε πρόβλημα σε κάποια πιο ευαίσθητα προϊόντα και γι' αυτό δεν περιλαμβάνεται αυτός ο παράγοντας στο τελικό πρότυπο γιατί δεν βρήκαν πολύ απλά στατιστική σχέση μεταξύ των δύο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις αυτές. Θα έχουμε μια συνεδρία οδόνες ηγητών ε, τις επόμενες ημέρες. Θα λάβετε λοιπόν τις δικές μας προτάσεις για ό,τι δεν μας ικανοποιεί απόλυτα μέχρι στιγμής και δεν καλύφθηκε από τις απαντήσεις. Ο κύριος Λούντι και από την Κομισιόν τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Θα εστιάσω σε κάποια βασικά σημεία που νομίζω ότι χρήζουν διευκρινήσεων. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το δίκτυο ε, το τεστ βελτίωσης ποιότητα, απαιτεί αύξηση στα επίπεδα υπηρεσιών, στο φάσμα των παρεχόμενων προ τον πελάτη προϊόντων και φυσικά αν υπάρχει ένα δίκτυο που προσφέρει ευρύτερη φάσμα υπηρεσιών στον πελάτη, αυτό σημαίνει και βελτίωση τη ποιότητα. Δεύτερο ερώτημα του εισηγητού για την καταγραφή των ε, τηλεφωνικών ε, αρχείων κτλ. Αν υπάρχει εκτέλεση παραγγελίας και αν έχουμε εκτέλεση μιας παραγγελίας, ε, πραγματικά έχουμε record keeping, αλλιώ, όχι. Έχουμε το record keeping στο πλαίσιο της οργνωσής της εταιρείας, είναι όμως κάτι διαφορετικό από τα τηλεφωνικά αρχεία. Τώρα, τα διαφορετικά μοντέλα στα διαφορετικά κράτη-μέλη δεν νομίζουμε ότι απέχουν τόσο πολύ το ένα από το άλλο. Το βασικό θεμελιώδη ζήτημα είναι να ληφθεί απόφαση μεταξύ διαχειριστή χαρτοφυλακίου και μεσίτη, ε, χρηματομεσίτη για την εκτέλεση μιας εμπορική συναλλαγής και την καταβολή κάποιων ε, αμοιβών για την έρευνα. Και σε ό,τι αφορά τι οργανωτικέ απαιτήσει, πρέπει να υπάρχει ένα λογαριασμό και ένα προπολογισμό. Και νομίζω ότι αν αυτό ισχύει, μπορεί να διατηρηθεί το CSA. Στην πράξη, τι μπορεί να γίνει. Εσωτερική έλεγχη εν μέρη και κάποιε ασφαλιστικέ δικλείδε των εταιριών θα πρέπει να επικαιροποιηθούν. Να έχουμε τον λογαριασμό πληρωμής έρευνα και διαφάνεια. Ποιο πληρώνεται γιατί. Και κατανομή στους διάφορους πελάτες. Με βάση την προκατρακτική μας ανάλυση, το θέμα δεν είναι τόσο ότι τα διαφορετικά κρατημέλη έχουν διαφορετικές απαιτήσει ό,τι αφορά τις προμήθειες αλλά είναι οι εταιρείε που θα πρέπει να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους για να υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους πόρους που δαπανούν. Για σε σχέση με του πελατές για του στόχου, πράγματι είναι δύο τα επίπεδα στόχευση αγοράς από τον κατασκευαστή και υποχρέωση του διανομέα να πωλεί σε πελάτες μέσα στη ορισμένη αγορά στόχο και δυνατόν μια ανάλυση πιο λεπτομεριακή των ομάδων στόχων με βάση τις παραμέτρους του κατασκευαστή για το συνολικό στόχο. Σε ό,τι αφορά τους ε, systemic internalizers. Ε, έχουμε εξετάσει 5, το κατόφλι των 5 εκατομμυρίων και ζητήσαμε νομική συμβουλή. Η ουσιαστική βάση όμως δεν μπορεί να οριστεί ε, έτσι περαιτέρω με, το, με μια κατεξουσιοδότηση πράξη. Πρέπει να σας πω ότι πολλοί διαπραγμάτες, πολλές συναλλαγές, ε, λιγότερο στοπίσιμα στοιχεία, ακόμη και στους systemic internalizers, ε, δεν υπόκειται στην υποχρέωση ε, της διαφάνειας πριν τη διαπραγμάτευση. Προπόθεση να υπάρχει διαπραγμάτευση τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα. Και ο τζίρο, ο ονομαστικό, να είναι συγκεκριμένο την μέρα. Και υπάρχουν κάποιε εταιρείε που θα είχαν αυτή την εξαίρεση των 5 εκατομμύρων, αλλά τελικά αποφελούνται από τις διάφορες απαιτήσει εφόσον μόνο στις αυτοποιήσιμες αγορές εφαρμόζεται η διαφάνεια. Uh, I want to briefly touch upon, ε, κάτι πολύ εύστοχο και το έχουμε μιλητήσει και εμείς, δηλαδή η ταξινόμηση ενός SI. Όταν έχουμε μία κατηγορία παραγωγονής SI για όλα τα ε, παράγωγα αυτή τη ε, τάξη, αυτή τη κατηγορία. Εμεί θεωρούμε ότι το πλαίσιο διαφάνεια, το RTS2 είναι το πλαίσιο και το κριτήριο. Έχουμε υποκατηγορίε παραγώγων με σόπς και πάρα πολλά άλλα αναλυτικά. Πολύ ε, λεπτομεριακά στοιχεία. Για το RTS2 κυρία Σουίνμπορν το ανέφερε. Πιστεύουμε ότι τα βασικά βήματα είναι η συμπερίληψη στα διάφορα στάδια του RTS. RTS είναι το, η βάση. Όμως έχουμε πει ότι προηγείται η έκθεση του RTS, αντίστροφα με ό,τι μέχρι τώρα. αν έχουμε καλούς όγκους διαπραγμάτευσης και όλα πηγαίνουν καλά, μετά πάμε στο επόμενο RTS. Περιμένουμε και στην τελευταία ε, εκδοχή του RTS ε, που εγκρίθηκε, θα ακολουθεί την ίδια προσέγγιση. Εμείς με το buy side έχουμε επαφές για την κατάρτιση του RTS Έχουμε έρθει σε επαφέ σε τακτά διαστηματά και πολλά από τα στοιχεία που τροφοδότησαν την ανάλυση μας ε, για το rds 2 Μα τα έδωσε το by side. Παρεπόμενες τώρα δραστηριότητες, πιστεύουμε ότι ένα κριτήριο είναι ε, το capital allocation. Μεταξύ των διαπραγμάτευσης και κρατοσκοπής διαπραγμάτευσης, αντίθεση με τις βασικές διαπραγματευτικέ ε, λοιπόν, δραστηριότητε και το capital allocation εκεί είναι ένα δύσκολο τεστ. Αλλά επειδή είμαστε στο επίπεδο 1 και επειδή οι νομοθέτε αποφάσισαν το κεφάλαιο e είναι ένα σχετικό κριτήριο, θα πρέπει να ορίσουμε ένα κατάλληλο τεστ και θα κάνουμε πάντο δυνατόν. Θα έχουμε διαβουλεύσει με του εμπλεκομένου φορεί για να επιλέξουμε το κατάλληλο από όλε τι επιλογέ που έχουν υποβληθεί από την ΕΣΜΑ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο. Είπαμε ότι την, έχουμε τη συνεδρία και μετά την Τρίτη. Την επόμενη Τρίτη το μεσημέρι που θα συζητήσουμε τα επόμενα βήματα και θα έχουμε ε, ίσως τότε λάβετε κάποια νέα αρτίες. Θα τα συζητήσουμε και αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μάιο και το προσωπικό του και τον ε, πρόσωπο της Κομισιόν και περνάμε σε κοινή συζήτηση επί του σημείου 4 και του σημείου 5 της ημερήσιας διάταξη σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα του κοινού κανόνε για την τιτλοποίηση και θέση του ευρωπαϊκού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση αφενό και για τι απαιτήσει προληπτική εποπτεία για πιστοτικά ιδρύματα και επιχειρήσει επενδύσεων αφετέρου. Προτείνω να ξεκινήσουμε με τον εισηγητή Πολ Τάν και του σκιώδη τη δική του έκθεση και μετά θα περάσουμε στον εισηγητή τη άλλη έκθεση, τον Πάμπλο, τον Πάμπλο Θάλβα και του σκιώδη του. Και από εκεί πέρα, αν έχουμε χρόνο, θα δώσω το λόγο και σε άλλου ομιλητέ. Θέλω όμω να σα υπενθυμίσω ότι επειδή έχουμε ένα πολύ μεγάλο κατάλογο μιλητών, πρέπει να εστιάσετε παρακαλούμε στα μείζωνα ζητήματα. Γιατί 11 και 4 έχουμε κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Απασχόλησης. Θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες ανακατατάξεις. Ε, δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να, να ε, επιμηκύνουμε ιδιαίτερα αυτή τη διαδικασία. Ε, δεν θα συνεχίσω άλλο εγώ να μιλάω. Δίνω αμέσως τώρα στον Πολ Τάγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, να μην αναλώσω πάρα πολύ από το χρόνο μας. Να πω καταρχάς ότι αν πραγματικά θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε την αγορά τιτλοποίησης, τιτλοποιημένων προϊόντων, θα πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα και να εφαρμόσουμε τα διδάγματα από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε τι δικηβεύεται αλλά και για να έχουμε και την υποστήριξη του κοινού. Να έχουμε δηλαδή προϊόντα τα οποία δεν θα είναι πλέον τοξικά. Θα πρέπει να πείσουμε και τους εαυτούς μας, αλλά και το κοινό και τους Ευρωπαίους πολίτες. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουμε μία επικοδομητική και επικριτική στάση παράλληλα. Όντως θεωρώ ότι τα τιτλοποιημένα προϊόντα έχουν τη δυνατότητα θεωρητικά τουλάχιστον να συμβάλλουν στην οικονομία, να υποστηρίξουν έμεσα και άμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορούν όντω να συμβάλλουν στην οικονομική διαφοροποίηση, έτσι ώστε να μην καταλήγουμε στην Ευρώπη να εξαρτώμαστε μόνο από τις τράπεζες, αλλά μπορούμε να έχουμε και διαφορετικά χρηματοπιστωτικά μέσα και φορείς και θεωρώ ότι μια αγορά τυπλοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι ίδιοι δηλαδή χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να γίνουν πιο υγιείς, πιο σταθεροί. Μέχρι σήμερα όμως μόνο λόγια είχαμε πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τις θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις και για το λόγο αυτό ακριβώς στην έκθεσή μου θέτω δύο βασικούς στόχους προκειμένου όντω να αντλήσουμε και να εφαρμόσουμε τα διδάγματα του παρελθόντος. Ο πρώτος στόχος έχει να κάνει με το διτό πρόβλημα της ασύμμετρης ενημέρωσης. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των συμφερόντων. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό αποθετήριο δεδομένων τυπλοποίησης. Αυτό το συζητήσαμε και σε ακρόαση και θεωρώ ότι μπορούμε μέσω του αποθετηρίου αυτού να έχουμε διαθέσιμα δημόσια δεδομένα τα οποία θα ωφελήσουν τόσο τους επενδυτές όσο και τις αρχές προκειμένου να γνωρίσουν ακριβώς ποια είναι η τοποθέτηση των επενδυτών αυτών, οι βασικές προθέσεις των επενδυτών. Ένα τέτοιο ευρωπαϊκό αποθετήριο δεδομένων τυπλοποίησης θα είναι υπέρ και του ίδιου του κλάδου, ακριβώς επειδή θα υπάρχει ένα μόνο σημείο επαφής, ένα σημείο ενημέρωσης, όπου θα συγκεντρώνονται όλα αυτά τα δεδομένα. Στα πλαίσια της ευθυγράμμισης στην οποία αναφέρθηκα, δεν θα πρέπει εδώ πέρα να έχουμε οποιαδήποτε ασάφεια προ προς την απονομή των ευθυνών. Γι' αυτό ακριβώ λέω εδώ πέρα ότι θα πρέπει να έχουμε και φορεί πιστοποίηση, να γνωρίζουμε ακριβώ ποιο είναι ο τελικό υπεύθυνο. Η ευθύνη όμω αυτή θα πρέπει να βαρύνει και τι εποπτικέ αρχέ. Έχουμε πλειονότητα, πληθώρα ρυθμιστικών εποπτικών αρχών στα κράτη-μέλη και είναι ασαφέ αυτή τη στιγμή ποιο είναι ο τελικό υπεύθυνο. Εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε την κατάσταση αυτή και να δώσουμε έναν ηγετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Επίσης, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τις κυρώσεις, σαφείς κυρώσεις που θα πρέπει να επιβληθούν. Από την άλλη υπάρχουν σαφή κριτήρια όσον αφορά τις κυρώσεις αυτές. Τα κριτήρια αυτά λοιπόν θα πρέπει να αποσαφινιστούν έτσι ώστε να μην καταλήγουμε στην δυσάρεστη αυτή κατάσταση πολλών ασαφών κριτηρίων και σαφών κυρώσεων από την άλλη. Αυτό είναι ο πρώτο στόχο. Ο δεύτερο στόχο έχει να κάνει με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και πραγματικά λυπάμαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή τη δεν έδωσε τη δέουσα σημασία στο σημείο αυτό. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα υψηλότερο επίπεδο διατήρηση, το οποίο δεν θα οδηγήσει μόνο σε ευθυγράμμιση των συμφερόντων αλλά από την άλλη θα λειτουργήσει εναντίον οποιοδήποτε δεινού οικονομικού κύκλου σαν αυτούς που αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγουμε αυτό που είχε συμβεί στο παρελθόν. Ιδιαίτερη ενίσχυση και μεγέθυνση της χρηματοπιστωτικής αγοράς, την οποία θα πρέπει να διχειριστεί στη συνέχεια μια τραπεζική αγορά η οποία δεν έχει τις απαραίτητες δυνατότητες να σταματήσουν επίσης τα φαινόμενα σκιώδους τραπεζική. Είναι το άλλο ζήτημα το οποίο έχω θέσει στην έκθεσή μου. Πρέπει και εδώ πέρα να υπάρχει το κατάλληλο υποπτικό καθεστώ. Πρέπει να, εξαιρεθεί επίσης, ε, να εξαιρεθούν ορισμένες μορφές CDNs, betting on bettings, σύνθετων δηλαδή μορφών τυπλοποίησης και πρέπει να δούμε επίσης τι μπορούμε να κάνουμε με τα ABCPs. Οι τυπλοποιήσει ABCP θεωρούνται πλέον πιο ασφαλείς, αλλά πρέπει και εδώ πέρα να υπάρχει απαραίτητη μακροληπτική εποπτεία. Αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε μια αγορά τυπλοποίησεων, η οποία θα συμβάλλει στην πραγματική οικονομία, που θα συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα, τότε η αγορά αυτή θα πρέπει να λειτουργεί καλά και τις καλές περιόδους, αλλά και τις δύσκολες περιόδους. Πρέπει να υπάρχει το παρέτο επίπεδο ρευστότητας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ, Πολ. Λυπάμαι που πιέζω για το χρόνο. Το λόγο τώρα έχει ο Σκιώδης εισηγητής από το ΕΛ Κότμαρ Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόκειται για μια αρκετά καλή βάση για την συζήτηση που ακολουθεί. Και βεβαίως απαιτείται περαιτέρω συζήτηση αφενός ο εισηγητής πράγματι στο έγγραφό του ανέφερε πως χρειάζεται διαφάνεια και λογοδοσία κάτι το οποίο πράγματι αναφέρεται στην εκκλησία. αλλά πρέπει να βρεθεί σωστή ισορροπία μεταξύ της διαφάνειας και της λογοδοσίας και βεβαίως ε, του ευθύνης και ενός κινήτρου απόδοσης για την αγορά. Γι' αυτό και οι τόσες τροπολογίες. Δεύτερον, όσον αφορά τις συνθετικές τυπλοποιήσεις, ε, έχουμε νομίζω μια καλή βάση πλέον. Ε, μιλάμε για μια αύξηση η οποία θα φτάσει από 5% στο 20% κάτι το οποίο θα συζητήσουμε και την επόμενη εβδομάδα και βεβαίως μιλάμε για τα διδάγματα που πρέπει να αντλήσουμε από την κρίση υπήρχαν τιτλοποιήσεις οι οποίες υποστήριξαν θετικά την πραγματική οικονομία οπότε αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να θεωρήσουμε άχρηστα όλα όσα υπήρχαν και λειτουργήσαν σωστά μέχρι στιγμής. Πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση. Οπότε χαίρομαι για την συζήτηση αυτή που υπάρχει και θα υπάρξει με τις τροπολογίες και την αναζήτηση ε, συμβιβασμών για να μπορέσουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια θέση του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ Ότμαρ. Λοιπόν, που επικεντρωθήκε στα μεγάλα ζητήματα. Για το ECR ο Μόρτεν Μέσα Σμιτ δεν είναι εδώ, αλλά είναι εδώ πέρα ο Σαΐντ Καμάλ. Ευχαριστώ, Μόρτεν. Ο Μόρτεν απουσιάζει και μου ζήτησε να μεταφέρω τα όσα έχει σημειώσει. Πρώτα απ' όλα λέει ότι υπάρχουν κομμάτια της έκθεσης που καλωσορίζει η ομάδα μας όσον αφορά την συνθετική τιτλοποίηση και τον αποκλεισμό κάθε είδους άρμπιτραζ από τα κριτήρια της ε, απλής ε, και διάφανης ε, τιτλοποίησης, αλλά θεωρεί πως θα πρέπει να υπάρξει και μια διαφοροποίηση με βάση τον ισολογισμό να παρέχουν χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία και ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μου ζήτησε να θέσω αυτά τα ζητήματα, ειδικά όσον αφορά την διακράτηση κινδύνου. Θεωρεί πως είχαμε συζητήσει τα ζητήματα στην προηγούμενη, στην ακρόαση της προηγούμενης εβδομάδας, στην οποία δυστυχώς απουσιάζαμε και οι δύο. Και η αύξηση της διακράτησης στο 20% ακριβώς δείχνει μια απόκληση από τα διεθνή κριτήρια και άρα θεωρεί πως πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω και αυτή τη στιγμή δεν βλέπει κάποια πιεστική ανάγκη για κάτι τέτοιο. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι επιπρόσθετες απαιτήσει διαφάνειας, έχοντας λάβει πολλές αντιδράσεις από ενδιαφερόμενους εκφράζουν αυτοί ανησυχίες για το κατά πόσον θα μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτές οι απαιτήσεις και δεν είναι σαφώς πως θα πρέπει να συμμορφωθούν οι διάφοροι φορείς. Επίσης υπάρχει ανησυχία πως ε, οι πληροφορίες όσον αφορά τους πραγματικούς ιδιοκτήτες ίσως ε, να ε, πηγαίνουν αντίθετα με την λειτουργία διαφόρων αποθετηρίων. Οπότε θα πρέπει πράγματι να επενδύσουμε επενδυτέ ε, στην αγορά τη τιτλοποίηση. Όσον αφορά αυτό το αποθετήριο δεδομένων, όπω είπαμε, το ECR έχει κάποιες επιφυλάξεις για άλλο ένα ευρωπαϊκό δημόσιο αρχείο, αλλά η επιλογή της Κομισιόν, όπου θα έχουμε πληροφορίες με βάση ένα τυποποιημένο υπόδειγμα, είναι επαρκής. Επίσης υπάρχουν οι συστάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας και υπό αυτό το πλαίσιο ε, επιτρέπεται η επανατιτλοποίηση αλλά υποκαθιστός υψηλότερων ε, χρεώσεων. Θα θέλαμε να το δούμε αυτό με τους γεωδησηγητές για τις ε, τρίτες χώρες. Θεωρεί πως οι τροπολογίες θέτουν το ζήτημα του εάν θα μπορούσαν να επενδύσουν τρίτες χώρες χωρίς να πηγαίνουν μέσω εξουσιοδοτημένων ταμείων. Έτσι θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση οι εκδότες ε, τίτλων από τρίτες ε, χώρες ε, και έτσι θα είχαμε και υψηλότερη συγκέντρωση του κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μόρδεν λοιπόν θα ήθελε να βρει λύσεις ε, για κάποιες από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν ε, για το αξιόχρεο κάποιων ε, χρηματοπιστωτικών οργανισμών τρίτων χώρων. Σας ευχαριστώ, Σαΐντ, μια της φιλελεύθερους. Θα δώσω λόγο στον Πίτερ Γιατσίκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με κάποια από αυτά που είπε ο εισηγητής επί παραδείγματι για μεγαλύτερη διαφάνεια για το SDR που θα εξυπηρετεί την πραγματική οικονομία, ακρογωνίας λίθους του όλου πλαισίου, θα πρέπει η ακολουθούμενη προσέγγιση να διοχετεύει τα αναγκαία στην πραγματική οικονομία, χρειάζεται επαρκής εποπτεία, υπάρχει ανάγκη για σαφήνεια όσον αφορά την ερμηνεία των κριτηρίων STS Συμφωνώ λοιπόν ότι η ΕΣΜΑ θα πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο. Συμφωνώ με την προσέγγιση για την πιστοποίηση των τρίτων μερών, για την ευθύνη της πιστοποίησης που θα πρέπει να ανήκει σε εκείνον που εκδίδει τα χρόγραφα. Θα πρέπει όμως ε, να εξασφαλίσει σωστή διαδικασία. Όμως έχω κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την ε, έκθεση κυρίως όσον αφορά κάποια θέματα, νομίζω ότι πηγαίνει πολύ μακριά και αυτό ίσως τελικά να καταστήσει το σύστημα μη ελκυστικό για τους επενδυτές και για τους εκδότες των τίτλων. Αυτό αφορά και την κατακάτηση του κινδύνου. Νομίζω ότι το 20% δεν αρκεί και πρέπει να εφαρμόζεται σε όλη την τιτλοποίηση και όχι απλώς τα STS είναι κάτι που δεν οδηγεί στην ποικιλομορφία των πηγών. Οι τράπεζες πρέπει να κρατούν στον ισολογισμό, παρακατούν το 20% και η τιτλοποίηση πλέον δεν γίνεται ελκυστική για τους ασφαλιστές και ούτε για τους τελικούς χρήστες. Το 5% εν γέννη μας βρίσκει συμφώνους. Θα πρέπει να έχουμε ένα γενικό πρότυπο ώστε να έχουμε ανταγωνιστική αγορά τιτλοποίησεων στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το 5% παρακράτηση του κινδύνου εκεί πρέπει να βρισκόμαστε. Για τους εκδότες των τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να κλείσουμε αυτομάτως την πόρτα σε αυτούς θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο αποφυγής αυτού όσον αφορά την κατάθεση των στοιχείων. Ε, θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τα στοιχεία και δεν είμαστε κατά μέτρων για να εξασφαλίζουν αυτό στην αγορά τιτλοποιήσεως. Θα πρέπει να εξετάσουμε λεπτομερέστερα το πόσο επηρεάζει το κόστος και την εφαρμοσιμότητα του πλαισίου STS μαζί με τις άλλες προτάσεις της εκθέσεως που θα αυξήσουν το κόστος για εκείνους που εκδίδουν τους τίτλους όπως η συγκράτηση του κινδύνου, ε, η δημοσιοποίηση στοιχείων. Ε, μήπως τελικά να αυξηθεί το κόστος στο SDS δεν είναι τόσο ελκυστικό. Επαναλαμβάνω κατά κλείδι ότι είμαι θετικός όσον αφορά το πλαίσιο αυτό, SDS, και υπάρχουν θετικά στοιχεία στην έκθεση TAN όμως εξακολουθούν να περιέχονται στοιχεία τα οποία ίσως να θέτουν σε κίνδυνο το ολοπλαίσιο διότι μπορεί να χάσει την ελκυστικότητά του και το STS μπορεί να γίνει κάτι απομονωμένο. Πρέπει να το επεξεργαστούμε και να γίνει κάτι πιο ελκυστικό το STS. Ευχαριστώ πολύ για την ΚΟΕ. Ο Μιγκουέλ Βιέγκος δεν είναι εδώ, αλλά ο Φάμπιο μήπως θέλει να πει κάτι. Ο Φάμπιο ρημάζει. Ε, ζητώ συγγνώμη από το σκιώδη του Μιγγέλ Βέκας που δεν μπορεί να είναι εδώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ε, πρότασή του. Ξεκινώντας από γενικά σχόλια, η πολιτική μου ομάδα επικρίνει το ολοπλαίσιο του STS, όπως δεν θα σε εκπλήσει αυτό. Ε, δεν είναι τυχαίο, ότι τελικά υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις το θέμα και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τα διάφορα χρηματοσυντικά συστήματα που χρησιμοποιούμε. Θα ήθελα να τονίσω λοιπόν ότι η πρώτη ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πετυχαίνει τον δηλωθέντα στόχο, δηλαδή τη βελτίωση της δανειοδοτήσεως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε όλες τους, τους, τις έρευνες κύρους όπως της Ευρωπαϊκής είδαμε ότι βασικό πρόβλημα των μικρομεσών επιχειρήσεων δεν είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αλλά η ζήτηση και ο συγητής το αναφέρει αυτό στην έκθεσή του, λέγοντας ότι είναι πολύ απίθανο ε, να πετύχουμε καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της χρηματοδοτήσεως των μικρομεσών επιχειρήσεων. Πιστεύουμε ότι οι μικρομεσαίες εξα... από καλά κεφαλοποιημένες ε, τράπεζες και από ζήτηση της αγοράς. Πάντα χρηματοδότηση ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν κάτι περιορισμένο όσον αφορά την αγορά τίτλων. Οι απαιτήσει για τη συγκράτηση του κινδύνου από 5 σε 20% είναι κάτι ευπρόσδεκτο. Η τροπολογία 48 μας προβληματίζει κάπως, όπου εκεί δημιουργείται μια εξαίρεση από τη βασική αρχή και πιστεύουμε ότι οι επενδυτές ε, για να μην επιτρέπουν να κάνουν επιλογή κινδύνων οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν μια ε, κάθετη μερίδα ε, και όχι μόνο οριζόντια μερίδα. Ε, στηρίζουμε και την αύξηση της διαφάνειας, κριτική απέτηση περί αυτού και η Financial Watch σήμερα το πρωί εξέδωσε μια ανακοίνωση σημαντική ακόμα και κατακαιρματισμένα στοιχεία είναι κάτι πολύ θολό για τους επενδυτές για να ενημερωθούν οπότε θα ε, βασίζονται σε εξωτερικούς αξιολογητές. Η Financial Watch έχει εκδώσει συγκεκριμένες ε, οδηγίες που θα θέλαμε να λάβει υπόψη η συγκητής. Υποστηρίζουμε την απαγόρευση της επανατιτλοποίησεως. Αναφέρθηκα στην πτυχή των διαφόρων κομματιών που δημιουργούνται. Πιστεύουμε ότι αναφορά σε, το, σε αναφορά των συνθετικών τίτλων σε ανέστιες θα πρέπει να αποφευθεί. Δεν το βρίσκουμε πολύ θετικό ως προσέγγιση αυτό που την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Φάμπιο. Για τους πράσινους δεν είναι εδώ Μόρις. Ο Σβένς Γκίργκολτ είναι εδώ όμως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μόλι κάνει εκστρατεία μέχρι την τελευταία στιγμή για να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε νομίζω δικαιολογείται. Θα διαβάσω τώρα την δήλωσή της και έχετε χαιρετίσματα. Σε γενικές γραμμές καλωσορίζουμε την επιφυλακτικότητα του εισηγητή για την απλή και διάφανη τίτλοποίηση και για το ποιο επωφελείται από την αναβίωση της τίτλοποίηση για να έχουμε αντλήσει τα διδάγματα από την κρίση. Εμείς θεωρούμε πως η πραγματική οικονομία αναζητεί δουλειές και όχι αυτόνομο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Θεωρούμε πω αυτοί οι οποίοι θα ωφεληθούν στην πραγματικότητα είναι η ενδιάμεση που θέλουν περισσότερη δραστηριότητα ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία και οι κεντρικές τράπεζες οι οποίες ε, βλέπουν ε, τους νέους τίτλους ε, ως απαραίτητους για την εντελώς ασυνήθιστη νομισματική πολιτική τους. Βλέπουμε εδώ πέρα πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να πάει παραπέρα από την Κομισιόν και το Συμβούλιο για να εστιάσει ακριβώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και να αντισταθεί στην πίεση για να υπάρξει μια αναδίπλωση όσον αφορά τις βελτιώσεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια. Σημαντικά σημεία εδώ πέρα είναι η διακράτηση κινδύνου κατά 20% αντί για το 5% που προτείνει η Κομισιόν και Συμβούλιο στο άρθρο 4,1 η απαγόρευση της επανατιτλοποίησης στο άρθρο 5β και ο περιορισμός στο τι μπορεί να είναι το υποκείμενο δάνειο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, σημείο 4. Επίσης υποστηρίζουμε μια νέα παράγραφο στο άρθρο 8.9 που απαγορεύει το αρμπιτράζ, τη συνθετική τιτλοποίηση από την ετικέτα απλής και διάφανης τιτλοποίησης. Η διαφάνεια δεν θα πρέπει να αφορά μόνο την τυπλοποίηση στο άρθρο 5 εδάφιο 1 και στον περιορισμό της αγοράς σε θεσμικούς επενδυτές ε, και ρυθμιζόμενες οντότητες στο άρθρο 2.8. Τέλος, στηρίζουμε τον ρόλο της ΕΣΜΑ και των εθνικών αρμοδίων αρχών έτσι ώστε να πληρούνται τα κριτήρια της απλής και διάφανης τυπλοποίησης Στο άρθρο 3α3 νέο και στην έκθεση της ΕΣΜΑ και στο άρθρο 5.1α. Επανερχόμαστε στο στην αρχή μας θέση ότι πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτά την πραγματική οικονομία και χαιρόμαστε για το άρθρο 10.3, μια νέα παράγραφο που έχει εκεί πέρα, που ζητάει να δούμε ποια θα είναι η επίπτωση στην πραγματική οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία γενικώ. Έχουμε όμως κάποιες επιφυλάξεις που ελπίζουμε ότι θα συζητηθούν υπό τον εισηγητή. Πρώτα απ' όλα η διατήρηση της αυτοπιστοποίησης, το άρθρο 14. Δεν ζητάμε από τους συμβαλόμενους να βεβαιώσουν την εγκυρότητα μιας σύμβασης. Είναι οι δικηγόροι ως ανεξάρτητοι ως ανεξάρτητα τρίτα μέρη. Το ίδιο και για την απλή και διάφαντη τυλοποίηση πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα το κάνει. Θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον η ανάγκη ευνηδιαστικών δειγματοληπτικών ελέγχων. Και επιπλέον, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θεωρούμε πω για να λειτουργήσει το σύστημα, η ποινή για λάθος ετικετοθεσία θα πρέπει να είναι αποτρεπτική. Είναι αφελές να θεωρούμε πω όσον οι αγοραστέ και οι πολιτέ είναι διατεθειμένοι να πιστοποιήσουν κάτι, ε, αυτό αρκεί. Έχουμε σοβαρές ανησυχίες για αυτό το οποίο λέει ο εισηγητής ότι δηλαδή θα πρέπει να περιληφθούν στην απλή και διάφανη τίτλοποίηση κάποιες συνθετικές τίτλοποιήσεις στο άρθρο 29 σημείο 3β. Η γραμμή μεταξύ αρμπιτράζ και ισολογισμών μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη για να την διακρίνει ακόμα και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Μας έχουν πει πως κάποια ασφάλιση πιστώσεων θα μπορούσε να θεωρηθεί συνθετική τιτλοποίηση. Η διάκριση πρέπει να είναι μεταξύ καλή την πίστη και μη ε, μεταβιβάσιμης ε, ασφάλειας και λοιπόν συνθετικών τιτλοποιήσεων. Θα θέλαμε λοιπόν να περιληφθούν και κάποια άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, Η ε, εποχικότητα θα συντομεύω γιατί βλέπω και πόσο ο πρόεδρος έχει δίκιο τελείωσαν τα πέντε λεπτά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα άρα θα τα υποβάλουμε στις ε, τροπολογίες μας. Θα ήθελα τέλος να πω πως η μη ευθυγράμμιση με το 5% της ε, ε, διακράτησης δεν ισχύει μόνο για την απλή και διάφανη τυλοποίηση, αλλά και για το παλαιό πλαίσιο της τυλοποίησης και θα χρησιμοποιήσουμε τον κανονισμό να, για να επαναφέρουμε όπως είπαμε, το θέμα αυτό της μη ευθυγράμμισης ε, για όλες τις τυκλοποίησεις. Ευχαριστώ. Η FTD Μάρκο Τζάνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την πρότασή του που λαμβάνει υπόψη κάποια σημεία προβληματικά που εξεφράστησαν και από τις ομάδες πολιτικές και από την κοινωνία των πολιτών όμως η θέση της ομάδας μου παραμένει άκρος επικριτική όσον αφορά την πρόταση αυτή για ένα βασικό λόγο. Είναι μια πρόταση που εν πάση περιπτώσει δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει στην επίλυση των προβλημάτων ε, που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στατιστικά στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική μιλούν καθαρά. Το πρώτο πρόβλημα για τι επιχειρήσει σήμερα δεν είναι η πρόσβαση στην πίστοση και στη ρευστότητα που παρουσιάζεται άφθονη ε, στο σύστημα στα πλαίσια νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, αλλά η έλλειψη ζήτησης είναι το πρόβλημα. Άρα αφετηρία για μας είναι ότι δεν θα αλλάξει τα πράγματα η πρόταση αυτής της επιχειρήσεις. Η μόνη θετική πλευρά που διαβλέπω είναι κάποια τέτοια στιγμή ε, μεγάλων ε, προβλημάτων για τους προϋπολογισμούς ε, και για τις τράπεζες. Αυτό μπορεί να είναι μια πρόταση, μπορεί να δημιουργήσει μια νέα αγορά, να αυξήσει το κεφάλαιο των αγορών. Αλλά αυτό που θέλουμε, το ερώτημα θέσουμε σε ποιο τίμημα, να αυξηθεί ο κίνδυνος, ο συστημικός κίνδυνος και εργαζόμεθα αντίθετα προς αυτή την κατεύθυνση και θα ήταν κρίμα. Εκείνος που επενδύει σε αυτού του είδους τα μέσα, οι θεσμικοί επενδυτές, του υπήν, που αναφέρονται στην έκθεση, είναι επενδυτές ε, οι οποίοι ήδη είναι πολύ στενά συνδεμένοι με το τραπεζικό σύστημα, κυρίως μέσω των διαφόρων συναλλαγών ρέπο και ρέπο markets. Με αυτή την πρόταση λοιπόν διακινδυνεύουμε να αυξήσουμε ε, το συστημικό κινδύνο, το συσχετισμό, δημιουργώντας αστάθεια μεγαλύτερη εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Άλλο σφάλμα που διαπράτεται κατά την άποψή μου είναι το εξή. Το να παίρνουμε προτάσεις που λειτουργούν σε άλλα συστήματα και να θεωρούμε ότι αυτές μπορούν να επαναληφθούν σε ένα σύστημα διαφορετικό όπως είναι αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την ε, είναι πολύ διαφορετική η Ευρώπη από τη ΣΥΠΑ εν γέννη. Όσον αφορά την χρήση των κεφαλαγορών, γνωρίζουμε ότι σήμερα στην Ευρώπη υπάρχει μια αγορά πολύ μεγάλη για ένα των cover bonds που είναι παρόμοιο την τοπίση παρόλο που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο προϊόντων. Ε, δεν νομίζω ότι τα STS μπορούν να αντικαταστήσουν αυτήν την αγορά που σήμερα οι τράπεζες και οι επενδυτές ε, προτιμούν όσον αφορά ε, αυτό το είδος ε, των στόχων. Όσον αφορά την ανεπάρκεια της προτάσεως αυτής, την αναποτελεσματικότητα, είναι πολύ ευρία η πρόταση και εδράζεται επί του κόστους. Αν καταφέρναμε να πετύχουμε τι έχουμε μέσω του STS ε, μία πρόταση στεναρή, συγκεκριμένη για διαφάνεια, για ε, και να υπάρχει σωστή πληροφορία που δίνεται, να υπάρχει συμμετρία στις χορηγούμενες πληροφορίες, τότε θα νικούσαμε δημιουργώντας ίσως ένα πλαίσιο για αυτού του είδους τα προϊόντα αποτελεσματικότερα. Την άλλη πλευρά όμως πιστεύω ότι αυτού του είδους το μέσο και αυτού του είδους η αγορά ε, δεν θα ακολουθεί το από τους φορείς αγοράς και της τράπεζας διότι το κόστος για να παραχθούν οι πληροφορίες για τον έλεγχο ε, τα underlying assets για να δώσουμε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες θα είναι πολύ μεγάλο οπότε θα είχαμε μια αγορά που δεν θα ήταν ε, ενδιαφέρουσα για τις τράπεζες. Επαναλαμβάνω λοιπόν για μια ακόμη φορά Λυπούμε διότι μεγάλες προσπάθειες που καταβάλουν οι πολιτικές ομάδες και που έκανε και ο εισηγητής δυστυχώς λίγο θα χρησιμεύσουν να πετύχουν το στόχο. Αυτό που χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα εργαστούμε, θα τονίσουμε τα σημεία μας, θα ενημερώσουμε τον συγητή, ευχαριστούμε τον συγητή για αυτά που έκανε όσον αφορά τη συγκράτηση του, του κινδύνου, το risk retention στο 20% είναι θετική η τοποθέτηση για το τελευταίο σημείο όσον αφορά τη συνθετική τιτλοποίηση και εμείς θα προτιμούσαμε ε, μια πλήρη απαγόρευση, ένα πλήρε μπαν αυτού του είδου των μέσων από το πλαίσιο του STS, διότι η χρήση παραγόγων ε, προϊόντων ε, νομίζω δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό του Simple Transparent Securization. Ευχαριστώ πολύ, Μάρκο. Δεν είναι εδώ Μπερνάρ μόνο. Πάμε στο σημείο 5 και μετά θα κάνω τελικό γύρο, αφού θα έχουν δυνατότητα να μιλήσουν τότε και άλλοι συναδελφοί. Ο Ο Πάμπλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και τώρα Θα μιλήσω ισπανικά. Νομίζω ότι συμφωνούμε σχεδόν όλοι τουλάχιστον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει σε μια πραγματική ένωση κεφαλαίου αγορών. Και ακριβώς η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης. Η Ένωση λοιπόν των Κεφαλαίων, η οποία κατά την άποψή μου θα πρέπει να βασίζεται σε δύο αρχές που θα επιτρέπουν στις χρηματαγορές να είναι πιο ολοκληρωμένες και ανοιχτές, ταυτόχρονα όμως και πιο ανταγωνιστικές και αποτελεσματικές. Αυτό αναμφίβολα θα ωφελήσει τους πάντες και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι ορισμένε ανησυχίε που εξέφρασαν και κάποιοι συνάδελφοι και στο πλαίσιο της έκθεσής μου είμαι διτεθειμένος να αναζητήσω λύσεις ε, ώστε οι ΜΜΕ να είναι πραγματικά αυτές που θα ωφεληθούν από μια τέτοια ένωση, της, ένωση των κεφαλαίων Ο συνάδελφος και εισηγητής ε, της άλλης έκθεσης για τις τετλοποιήσεις μας είπε ότι θα πρέπει να μας διδάξει πράγματα η κρίση και συμφωνώ. Πρέπει να είμαστε και ρεαλιστέ όμω, αλλά και να έχουμε επίγνωση ότι η χρηματοπιστωτική κρίση από το 2007 έω το 2008 ή τέλο πάντων μέχρι τότε μέχρι την κρίση οι χρηματαγορές, ε, οι χρηματοπιστωτικές αγορές ε, λειτουργούσαν ε, λογικά και είχαν και, αύξη, συνεχή ανάπτυξη. Και αυτό που είναι και πιο σημαντικό στη διάρκεια τη οικονομική κρίση. Αυτού του είδους τα προϊόντα είχαν λογικά καλά αποτελέσματα. Δηλαδή ήταν ελάχιστον σημασία οι απόλυες που είχαν. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτά τα προϊόντα έχουν μια καλή φήμη και καλό είναι να μην ε, χάσουν αυτή τη φήμη και να μην στιγματιστούν. Και ε, είναι ακόμα πιο μεγάλη ζημία λόγω ανεύθυνων συμπεριφορών ορισμένων ε, ανθρώπων για, μιλώ για άλλες περιοχές του κόσμου σε σχέση με αυτά τα πρώτα και κυρίως μιλώ για τη ΣΥΠΑ βέβαια. Ο Πολ Τάγκ μίλησε και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη αυτό το γεγονός. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε ποτέ, να, να επιτρέψουμε ποτέ να γυρίσουμε πίσω σε αυτό το αρνητικό παρελθόν. Και το έχουμε αυτό υπόψη μας ε, ως στόχο κατά τη σύνταξη των αλλά δεν ξεχνάμε ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να συνεισφέρουμε ώστε να επανέλθει και η βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, αυτέ πρέπει να είναι προτεραιότητε. Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα αφενό και ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη αφετέρου. Η διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότηση έχει για μένα κεφαλαιότητα σημασία στην ε, κεφάλαιο αγορά εδώ στην Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες για τους επενδυτές. Η χρηματοδότηση πρέπει να συνδεθεί με την πραγματική οικονομία. Πρέπει να προωθήσουμε για μια ακόμη φορά ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα είναι ενισχυμένο και πιο ανθεκτικό. Και πρέπει επίσης να εμβαθύνουμε στη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό. Με τη δημιουργία ενό μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά τιτλοποίηση ψηλή ποιότητα θα συνεισφέρουμε στην επίτευξη αυτών των στόχων και θα οδηγήσουμε σε μεγαλύτερη ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαστεί επίσης να διαφοροποιηθούν οι πηγές χρηματοδότησης και να δοθεί βοήθεια για την απεμπλοκή κεφαλαίων που δεν χρησιμοποιούνται επί του παρόντος. Άρα οι, οι δύο επιχειρήσεις αλλά και γενικά οι επιχειρήσεις δεν διευκολύνονται αυτή τη στιγμή. Αλλά θα πρέπει να το κάνουμε αυτό και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να πάρουν πιο εύκολα δάνειο. Έρχομαι λοιπόν σε κάποια στοιχεία της δικής μου έκθεσης. Μία από τις πτυχές που προτείνω να τροποποιηθεί είναι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Είναι σημαντικό να έχουμε τη σωστή ιεράρχηση, τη σωστή εστίαση για αυτό το νομοθετικό πακέτο. Η πρόταση του Συμβουλίου και η πρόταση της Κομισιόν συνιστούν σημαντικά βήματα προς τη δημιουργία ισότητας ευκαιριών και συνθήκων στην ε, Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Και θα πρέπει δίκαια να καθοριστούν οι διάφορες απαιτήσει, αλλά, οι κεφαλικές απαιτήσει, αλλά σε ό,τι αφορά τα external ratings, ε, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε εστίαση για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την αγορά και όχι να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη σύγκριση με τη ΣΥΠΑ. Η πρόταση αυτή ευθυγραμμίζεται και με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεύτερον, η Ένωση Κεφαλαίου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια ένωση που εστιάζει απόλυτα και αποκλειστικά στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους μεγάλους ομίλους. Το αντίθετο, θα έλεγα. Οι βασικοί δικαιούχοι και ωφελημένοι πρέπει να είναι οι επιχειρήσεις, που είναι και ο και η ατμομηχανή τη ανάπτυξης και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε στι μικρομεσαίε επιχειρήσει ένα πιο ευρύ φάσμα επιλογών για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν, να διαφοροποιήσουν τι πηγέ χρηματοδότησή του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο όπω μέχρι στιγμή ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό ίσχυε ε, από τις ε, τράπεζες που είναι κοντά στο, στην έδρα τους, αλλά θα μπορούσαν να εξεταστούν και άλλες επιλογές σε μια αγορά ανάπτυξη, επένδυση κεφαλαίου, που δεν θα προέρχεται μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες χώρες. Η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οποιαδήποτε υπόδειξη προς αυτή την κατεύθυνση του συναδέλφου μου θα ήταν κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη. Αυτά είχα να σας πω. Επαναλαμβάνω, οποιαδήποτε σχόλιο, οποιαδήποτε υπόδειξη και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ Παύλο. Θα περάσουμε απευθείας στους σκιώδης εισηγητές με πρώτον το σκιώδη Σοσιαλιστών Δημοκρατών, Γιώνας Φερνάνδη. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε, εδώ συζητάμε δύο εκθέσεις που υποτίθεται πρέπει να επηρεάσουν ξεκάθαρα ε, την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. για βελτίωση και της νομισματικής πολιτικής της ΣΕΚΤ, ε, αύξηση του τραπεζικού πολλαπλασιαστή. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τον ε, Παύλο Θάλμπα για την έκθεσή του. Πιστεύω ότι επισημαίνει ορισμένες γραμμές ε, τις οποίες θα πρέπει να τροποποιήσουμε με την νομοθετική διαδικασία Υπάρχουν βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και κάποιες διαφορές στις απόψεις μας. Πριν περάσω όμως στην ε, έκθεση Στάλβα, θέλω να πω ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση των κεφαλαικών απαιτήσεων θα μπορούσε να δεχθεί η ομάδα μας ε, για τις STS την απλή διάφανη τυποποιημένη τυπλοποίηση θα πρέπει να περνά από την έκθεση Paul Tank και την τροποποίησή της. Επαναλαμβάνω, είμαστε διατεθειμένοι και αυτή είναι και δουλειά μας να διαπραγματευτούμε τις κεφαλαιακές απαιτήσει ε, για τις ε, τετλοποίησεις STS, απλές διάφανες και τυποποιημένες, όμως Υπάρχουν και άλλες τυπλοποίησει και το τι θα γίνει με αυτές αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς προχωρεί η διαπραγμάτευση της έκθεση του Πολ Τάγκ, ο ε, προτείνει μέτρα για μεγαλύτερη ασφάλεια και για την ε, δική μας ομάδα αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Όπως είπα λοιπόν, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για την έκθεση θα δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και τις κεφαλαιακές απαιτήσει που θα πρέπει να εφαρμόσουμε σε αυτές τις δηλοποίησεις STS. Τώρα, πέραν από τις αρχικές μου αυτές απόψεις, πρέπει να πω ότι η ομάδα μου θεωρεί ότι η και αξιολόγηση. δεν θα πρέπει να ξαναμπούν ε, στους σχετικούς ε, κανονισμούς και ρυθμίσεις. Είναι ένα από τα διδάγματα που αποκομίσαμε με την κρίση, ότι δηλαδή πρέπει να αποφύγουμε την ε, ανάμιξη αυτών των εικοναξιολόγησης και επομένως νομίζω ότι πρέπει όταν θα υπολογίζουμε τις κεφαλαϊκές απαιτήσει ε, για τα STS, δεν είναι καλή ιδέα να ξαναβάλουμε στο προσκήνιο της κοσαξιολόγηση. Συμφωνούμε ε, λοιπόν με την άποψη του εισηγητή και ελπίζουμε να υπάρξουν ε, ε λύσεις γιατί υπάρχουν εναλλακτικά συστήματα. Τώρα, στο βαθμό που θεωρούμε ότι η εστερική μέθοδος πρέπει να έχει περισσότερη βαρύτητα για τον υπολογισμό των κεφαλαίων απαιτήσεων, δεν συμφωνούμε με την πρόταση του εισηγητή για μείωση από το 95% στο 80% ε, των υποκείμενων πιστώσεων στις τιτλοποιήσεις ε, για να επιτρέπεται η χρήση του εσωτερικού μηχανισμού. Δεν πιστεύουμε ότι γίνεται να δεχθούμε συστήματα που δεν ξεκαθαρίζουν ε, ότι πρέπει να υπάρχει καλή ενημέρωση και διαφάνεια σε ό,τι αφορά ε, την πίστοση για να μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά αυτό το σύστημα. Από την άλλη πλευρά, έχουμε σοβαρές αμφιβολίες ως ομάδα σε ό,τι αφορά τι συνθετικέ επιλοποιησει ε, Τα εξήγησε ο Πολ Τάνκ ε, στην προηγούμενη έκθεση. Η πρόταση της Κομισιόν, από αυτήν την έννοια, διευρύνει ή τέλος πάντων επιτρέπει τη χρήση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις ε, συνθετικές τετλοποίησεις όταν υπάρχει ε, κάποια εγγύηση που παρέχεται από μια οργάνωση που έχουμε μηδενική έκδοση, δημόσιες τράπεζες, πολλές περιπτώσεις κτλ. Ο εισηγητής όμως διευρύνει το πεδίο για τη χρήση αυτών των ειδών ε, απαιτήσεων για τις συνθετικές τετριλοποιήσεις, ε, τα, ε, μιλάει για καταθέσεις σε μετρητό κτλ. Αυτή η ε, διεύρυνση για τη χρήση των για τη χρήση αυτών των ακεφαλαιοκών απαιτήσεων στις συνθετικές τυπλοποιήσεις είναι στα όρια αυτού που εμείς θα θεωρούσαμε σκόπιμο και θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις στην έκθεση του Πολ Τάνκ, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, σε σχέση με αυτές τις συνθετικές τυπλοποιήσεις. Σε ό,τι αφορά τη, τα δάνεια προς τις ΜΜΕ συμφωνούμε αυτό, το 80 προς 70% που μειώνεται η δυνατότητα χρήσης αυτών των ε, ελασσόνων απαιτήσεων ε, για τα PCB και για τις υποκείμενες πιστώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν ξέρω. Θέλουμε να διευκολύνουμε τη χορήγηση δανείων ε, στις ΜΜΕ, αλλά όχι να μειώνουμε αυτά τα ποσοστά, πρέπει να τα αυξήσουμε αντίθετα για να ωφεληθούν πράγματι οι ΜΜΕ και όχι άλλε επιχειρήσεις. Τέλος, θεωρούμε ότι υπάρχει μια φιλοσοφία πίσω από αυτήν την έκθεση, η οποία θα μπορούσε να ε, συμβαδίσει με τα όσα λέγω στην έκθεση του Πολ Τάγκ. Ευχαριστώ. Πρέπει να παραμένουμε όμω εντό του χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, είσαι Άρκε Σαΐτ Καμάλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα μιλήσω εξ ονόματός μου, αλλά και της ομάδας βεβαίω. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε τον Πάμπλο για τη δουλειά που έκανε και έφτιαξε κάποια σημαντικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα για την μέθοδο ιεράρχησης. Αντιλαμβανόμαστε το σκεπτικό του εισηγητή και όσον αφορά την αλλαγή της ιεραρχίας και τα επακόλουθα μοντέλα και έχετε δίκιο όσον αφορά την απλότητα, αλλά ε, δεδομένου του αντικειμένου δεν ξέρω αν ποτέ θα μπορέσουμε να έχουμε την απλότητα αυτή. Το ECR βεβαίω είναι υπέρ του στόχου της μείωσης του ρόλου των ε, οίκων και πράγματι εδώ πέρα προσπαθούμε να περιορίσουμε τις ασυνέπειες που υπάρχουν. Όμως κάποιοι ενδιαφερόμενοι έχουν εκφράσει ανησυχίες, ε, παραδείγματος χάρη ο κλάδος των δανείων για αυτοκίνητα έχουν πει πως και με τις τροπολογίες αυτές θα υποφέρουν αν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εξωτερική αυτή μέθοδο και πρέπει να το συζητήσουμε μαζί τους να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εσωτερική μέθοδο και αν μπορεί αυτή να εφαρμοστεί ή τους αυξάνει το κόστος ή δεν τους επιτρέπει να δουλέψουν. Μετά. έχουμε κάποιες ε, προσαρμογές στην μέθοδο της ε, εσωτερικής αξιολόγησης ε, και λέμε ότι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεδομένα τρίτων και θεωρούμε πως έτσι θα υπάρξει μια αντιστοιχεία μεγαλύτερη μεταξύ επενδυτών στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ανησυχούμε γιατί δεν είχαν επιτραπεί αυτές οι μέθοδοι στο παρελθόν και πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη σαφήνεια για το τι περιλαμβάνει αυτό και βεβαίως ε, και ποιον θα καλύπτει και σε ποιο βαθμό για τις ε, προσαρμογές στην τυποποιημένη προσέγγιση. Έχουμε το άρθρο 258, το νέο 258α που επιτρέπεται στις αρχές ε, να αποκλείσουν την χρήση αυτή. Και βεβαίως πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι STS σημαίνει απλή, διάφανη και τυποποιημένη ε, και πρέπει να μην χρησιμοποιούμε πάρα πολύ περίπλοκα μέσα και να μην επιτρέψουμε στον κλάδο να κάνει ό,τι θέλει. Καλώς ορίζουμε λοιπόν την αναγνώριση ότι πράγματι θα συνεχίσουν να υπάρχουν περίπλοκα προϊόντα που μην θα είναι απλά και τυποποιημένα, αλλά πρέπει να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα και βεβαίως αυτό είναι θέμα μεταξύ των εισηγητών του Πάμπλο και του κύριου Τάγκ ε, το πώς θα τα συντονίσουμε στο μέλλον. Δηλαδή τα απλά και διάφανα και τυποποιημένα και αυτά που δεν είναι τέτοια. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στους φιλελεύθερους. Ο Μάικλ Τόιρερ. Να ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήδη υπόθηκαν αρκετά και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και βεβαίως ε, ο Πέτερη Γέσεκ ε, εξέφρασε την ανησυχία πως ε, έχουμε όλο αυτό το πακέτο της τιτλοποίησης και μήπως μαζί με τα ξερά καούν και τα χλωρά γιατί η τιτλοποίηση στις ΕΠΑ έπαιξε μεγάλο ρόλο στην οικονομική κρίση όμως βλέπουμε πως υπάρχει μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση της κατάστασης ε, στην Ευρώπη και δεν ήταν ε, όλα επικριτικά. Αντιθέτως υπήρχαν κάποια προϊόντα τίτλοποίησης τα οποία δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα με την κρίση. Ήταν πάρα πολύ ασφαλή και σε αντίθεση με τα asset-backed securities ξέρουμε πάρα πολύ καλά το τι τίτλοποιείται. Οπότε τώρα το να υπάρξει μια απλή αύξηση της ε, στάθμισης του κινδύνου δεν σημαίνει ότι θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τον στόχο της αναζωογόνησης αυτής της αγοράς στην Ευρώπη. Κάποιες λεπτομέρειες αναφέρθηκαν ήδη και από τους ενδιαφερόμενους ε, που ζουν τα πράγματα καθημερινά. Σκεφτόμαστε λοιπόν ε, σε ποια σημεία θα μπορούσαμε να παρέμβουμε και να καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες. Θεωρούμε πως δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κενό, κάποια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ ε, της ε, αντιμετώπισης covered bonds και asset backed securities. Επιπλέον αναρωτιόμαστε εάν αυτά τα οποία προτείνει ο Παύλος Ζάλμπα, η αλλαγή δηλαδή ε, της ε, κατάταξης της ε, Κομισιόν μεταξύ IRBA, ERBA και STS ε, λύνει το πρόβλημα. Προσπαθούμε δηλαδή έτσι να βγάλουμε τους, τίτλους, τους οίκους αξιολόγησης ε, από την τίτλοποίηση. Εδώ πέρα αμφιβάλλουμε γιατί ειδικά τα asset-backed ε, commercial papers θα επηρεαστούν αρνητικά. Και μέχρι στιγμής ε, ούτε η ΕΣΜΑ ούτε η Κομισιόν έχει προτείνει κάποια λύση. Εμείς θα θέλαμε τα asset-backed commercial papers και στο μέλλον να συνεχίσουν να εφίστανται γιατί εξαρτά, εξαρτά, εξαρτάται από αυτά η πραγματική οικονομία. Είτε μιλάμε για δάνεια για αυτοκίνητα, είτε για μηχανολογικό εξοπλισμό και την ε, μισθωσή του το θέμα της ε, τίτλοποίησης, ε, εάν απαγορευτεί σε αυτόν τον κλάδο, θα επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά την πραγματική οικονομία. Λοιπόν, τα asset-backed commercial papers, ε, όπως είπα, περιέχουν σοβαρούς κινδύνους γιατί είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την πραγματική οικονομία. Οπότε θεωρώ πως εδώ πέρα θα πρέπει να αναλύσουμε προσεκτικά και από κοινού το πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε να αποκλείσουμε τα asset commercial papers και θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε και την προσέγγιση της εσωτερικής αξιολόγησης που θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον. Ε, βεβαίως θα πρέπει όπως είπαμε να ξανακινηθεί η σχετική αγορά στην Ευρώπη, κάτι το οποίο υποστηρίζει η ομάδα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στην Γκουε. Εσείς ε, λοιπόν αντικαθιστάτε τους πάντες. Φάμπιο Ντεμάζη λοιπόν πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ τον Παύλο Ζάλμπα για την ε, πρότασή του. Ανέφερα την γενική μας άποψη για το θέμα της ε, τηλεοποίησης σε αντίθεση με τα όσα είπε ο Πάμπλο. Εμείς δεν βλέπουμε σοβαρά στοιχεία για την σύνδεση της ε, μεθόδου αυτής χρηματοδότησης με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, το αποδεικνύουν, αλλά επειδή ο Μάικλ είπε ότι ε, δεν θα είχαμε τα ίδια προβλήματα στην Ευρώπη. Θα ήθελα να πω πως όταν ξέσπασε η κρίση της ΕΠΑ, κάποιες χώρες όπως η Γαλλία ήταν έτοιμες να απελευθερώσουν το νομικό πλαίσιο για αυτές τις δραστηριότητες, οπότε εάν αν περιμέναμε ένα-δύο χρόνια ακόμα θα είχαμε τα ίδια προβλήματα και εδώ. Όμως, Θεωρώ πως ο πραγματικός στόχος της πρότασης αυτής είναι να ξεφορτωθούν οι τράπεζες κάποια στοιχεία του ενεργητικού τους. Ε, να το κάνουν, αλλά το θέμα είναι πώς. Εμείς δεν θεωρούμε ότι με το να τα πασάρουν στην υπόλοιπη κοινωνία θα γίνει πιο σταθερό το τραπεζικό σύστημα. Τέλος πάντων, στη συγκεκριμένη έκθεση τρία σχόλια. Θεωρούμε πως ο εισηγητής ε, έχει κάποια αρνητική θέση και που τροποποιεί την πρόταση της Κομισιόν. και όπου λέει ότι η προσέγγιση της εσωτερικής αξιολόγησης πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της ε, τυποποιημένης ε, προσέγγισης γιατί βλέπουμε ότι σε παρόμοια στοιχεία δίνουν τελείω διαφορετική αξιολόγηση οι τράπεζε. και είμαστε επιφυλακτικοί για το ότι προτείνει ο Συγητή να χαμηλώσουν οι ελάχιστε απαιτήσει για την εσωτερική αξιολόγηση κινδύνου. Σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει η Κομισιόν θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα 95% του ποσού της έκθεσης, το οποίο θα αποτελέσει βάση, εδώ πέρα προτείνεται να το κατεβάσουμε στο 80% και δεν αναφέρεστε σε αυτό το οποίο λέει η Κομισιόν το να ανέβει το κατέφλι στο 10%. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανέβει πολύ περισσότερο. Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε για την ε, πρόταση και ελπίζω να έχουμε μια καλή συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον από τους πράσινους. Σβέν. Δεν αντικαθιστάς κάποιον. Ωραία. Λοιπόν, Μάρκο Βάλλη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχά κάποιες γενικές παρατηρήσεις πολιτικής φύσης. Ως πολιτική ομάδα είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί, όπως το είπα και προηγούμενα, για την πρόταση αυτή τιτλοποίησης, για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και την πρόταση του εισηγητή. Θεωρούμε ότι δεν βοηθούν οι προτάσεις αυτές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αντίθετα υπάρχουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι αύξηση του συστημικού κινδύνου, ότι μπορεί να δημιουργηθεί νέα φούσκα όσον αφορά τα ακίνητα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να διαχειριστούμε τα έσοδα των τραπεζών με τον πιο διαφανή δυνατό τρόπο. Επίσης έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη αυτή πρόταση ακριβώς επειδή ελοχεύουν πολύ συστημικοί κίνδυνη. Θα προτιμούσαμε να μπορούσαμε μέσω των πολιτικών μας αποφάσεων να περιορίσουμε τους κινδύνους αυτούς και νομίζω ότι ακριβώς αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να περιχαράξουμε το σύστημα αυτό για να περιορίσουμε τους κινδύνους, αλλά δυστυχώς δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι χρειάζεται επίση και ένα σοβαρό σχέδιο δημοσίων επενδύσεων. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα πάρει πάλι μπρο η οικονομία. Αλλά φαίνεται το ζήτημα αυτό είναι ταμπού, κανεί δεν θέλει να το θίξει. Και Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι οι λύσεις που προτείνονται τελικά δεν βοηθούν πραγματικά την οικονομία, αλλά μόνο τις τράπεζες και το χρηματοπιστωτικό τομέα. Σε σχέση τώρα με την πρόταση του Πάμπλο, πάλι εδώ πέρα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες επικρίσεις όσον αφορά καταρχά τις απαιτήσει προληπτικής εποπτείας, Πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να το δούμε εδώ. Η συμπερίληψη των, της συνθετικής τιτλοποίησης, αναφερόμαστε εδώ πέρα σε παράγωγα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η διασύνδεση ανάμεσα στην πραγματική οικονομία και όλα αυτά τα προϊόντα τιτλο, Δεν ξέρω πραγματικά αν θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερες ε, αδειοδοτήσεις διαπραγμάτευσης στους εμπλεκομένους στο χρηματοπιστωτικό τομέα, οι οποίοι θα συνεχίζουν να παίζουν τελικά με όλα αυτά τα μέσα εις βάρος πραγματικής οικονομίας. Επίσης, εσωτερική ε, βαθμολόγηση και πάλι δεν είναι διαφανής εδώ πέρα η ε, διαδικασία. Όσον αφορά τις εξωτερικές διαβαθμίσεις, ως προς αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα λειτουργούν οι ε, οίκοι αξιολόγησης, να ακολουθούν συγκεκριμένη αμερόληπτη και διαφανή προσέγγιση, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δίνω τη δυνατότητα σε μια τράπεζα χρηματοπιστωτικό οργανισμό να αυτοπιστοποιείται, τα πράγματα δεν λειτουργούν θετικά. Επίσης, έχουμε διάφορες επιπτώσεις μόχλευσης στο χρηματοπιστωτικό τομέα, οι που οδηγούν σε συστημικά προβλήματα. Τώρα το να έχουμε σε ένα μοναδικό προϊόν διαφορετικά προφίλ κινδύνου και αυτό προτείνεται στην πρόταση. Μα με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε τελικά σύνθετα, ασαφή προϊόντα, τα οποία δεν είναι απλά και διαφανή, όπως ακριβώς υποτίθεται ότι είναι η πρόθεση της πρότασης αυτής. Από τη μια μιλάμε για μια πρόταση STS και μέσα στην πρόταση αυτή κρύβονται τελικά προϊόντα τα οποία δεν είναι διαφανή είναι τυποποιημένα σίγουρα, αλλά σίγουρα δεν είναι ούτε απλά ούτε διαφανή. Υπάρχει λοιπόν μια σημαντική αντίφαση στο σημείο αυτό και είμαι στη θεσή σα για να κάνουμε και περαιτέρω προτάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλει κανεί άλλο το λόγο. Όχι, μάλλον κάποιος θέλει το λόγο, συγγνώμη. Να ακούσουμε λοιπόν κάποιου ομιλητέ ακόμα πρωτού κλείσει ο κατάλογο των ομιλητών. Νίνα Γκίλ, παρακαλώ. Ο Πολ και ο Παύλο μετά. Ευχαριστώ. Να συγχαρώ καταρχά τον συνάδελφό μου τον Πολ για, το φωτο, για αυτό το σχέδιο έκθεση, το οποίο θεωρώ ότι είναι μια φιλόδοξη έκθεση που πετυχαίνει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην αναζωογονοποίηση τη αγορά τυπλοποίηση και την τόνωση της πραγματική οικονομίας. Νομίζω όμω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχουν και απαραίτητε εγγύησει για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ότι θα πρέπει να δίνονται και οι απαραίτητε διασφαλίσει ενημέρωση και πληροφόρηση. Είναι σημαντικό σαφώ να μην επιστρέψουμε σε προηγούμενε καταστάσει, σαφώ να αντλήσουμε τα διδάγματα του παρελθόντο και ω προ αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε καλύτερη εποπτεία. Ποιο είναι το ρίσκ κινδύνου, τι ακριβώ τυπλοποιείται και παράλληλα θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος επενδύει τελικά στα τιτλοποιημένα αυτά προϊόντα. Μέχρι σήμερα όλα αυτά δεν ήταν ιδιαίτερα σαφή, ήταν μάλλον ασαφείς και κρυφές διαδικασίες. Αν πραγματικά λοιπόν τα STS θέλουμε να είναι πιο ασφαλή και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε περαιτέρω φούσκες και κερδοσκοπίες, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια σε όλο το εύρος της αγοράς τιτλοποιήσεων. Περισσότερο, λοιπόν να διαφάνει όπως ακριβώς ζήτησε και ο εισηγητής και αυτή είναι καθοριστική προϋπόθεση για τη δημιουργία απλών διαφανών και τυποποιημένων τυπλοποιήσεων. Πρέπει έπειτα να υπάρχει και απαραίτητη συνεργασία όσον αφορά τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Όσον αφορά αυτό το ευρωπαϊκό απόθεμα για τα προϊόντα τυπλοποίησης, σαφώς θα μπορούσε, το αποθετήριο με συγχωρείτε, σαφώς θα μπορούσε να μας βοηθήσει, αλλά πρέπει να λειτουργεί με το σωστό τρόπο. Και μια παρατήρηση ως προς αυτό. Θέλουμε αυτή τη στιγμή να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτός είναι ο πιο βασικός παράγοντας σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα τα πράγματα περιπλέκονται κάπως για τους επενδυτές εκείνους που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η άποψη του Πολ ως προς αυτό. Ενδεχομένως κάποια από τα πράγματα προτείνονται εδώ πέρα να δημιουργούν προβλήματα στους ξένους επενδυτές. Επίσης, για να λειτουργήσει καλά αυτό το ευρωπαϊκό αποθετήριο δεδομένων τυπλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφώς ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό. Ίσως και η ΕΣΜΑ θα μπορούσε εδώ πέρα να διδραματίσει κάποιο ρόλο. Μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού του αποθετηρίου, αλλά όχι να έχει την πλήρη διαχείρισή του. Ευχαριστούμε πολύ, Νίνα. Καταρχάς τώρα το λόγο έχει ο Πολ Τάν και στη συνέχεια ο Παύλο Θάλμπα. Πόλ. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Θα, Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση. Πολλά θέματα έχουν φυγεί. Βλέπω όμως ότι υπάρχει μια ευρεία συμφωνία. Χρειαζόμαστε διαφάνεια, λογοδοσία ταυτόχρονα. Αυτές είναι σημαντικές αρχές που πρέπει να επεξεργαστούμε. Μετά υπάρχουν ανησυχίες για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα αναφέρθηκε το πρόβλημα του συστημικού κινδύνου και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό. Βλέπω ότι στο Κοινοβούλιο συζητούμε τα ίδια θέματα, έχουμε διαφορές, αλλά σε γενικές γραμμές συμφωνούμε επί των διαφόρων αρχών. Και αυτό είναι θετικό. Πολλά θέματα πρέπει να εξεταστούν πώς θα λειτουργήσει η διαφάνεια αναλογικά. Αυτό είναι ένα καλό θέμα συζητήσεως, αλλά και αυτό που είπε η Νίνα, πώς συμπεριλαμβάνουμε τρίτες χώρες, διότι υποθέτω ε, δεν θα υπάρχει τίτλος απλούς και, απλής και διαφανής ε, διαδικασίας, απλού και διαφανούς τίτλου, πώς θα έχουμε τις σωστές συναλλαγές με τρίτες χώρες. Πρέπει να το επεξεργαστούμε αυτό. Μετά από τις συζητήσεις ε, προσβλέπω σε μελλοντική κουβέντα διότι βλέπω ότι ακολουθήθηκε και κριτική προσέγγιση αλλά και επικοδομητική και αυτό αποτελεί μια καλή αφαιρετήρια. Ευχαριστώ πολύ Πολ για Ο Πάμπλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους τους συναδέλφους ε, για τα σχόλιά τους που είναι όλα επικοδομητικά. Θα κάνω σχόλια για παράδειγμα, σε σχέση με τον κύριο Χώνας Φερνάντεθ για την ε, νομισματική πολιτική, είναι κοινό ο στόχος μας και ελπίζω με αυτές τις εκθέσεις ε, να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, να βελτιώσουμε τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Στόχος βέβαια και πεδίο εφαρμογής έκθεση δεν είναι η Ευρωζώνη μόνο, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Βέβαια, Κάποιες αγορές, ε, ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές σίγουρα θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη με τις νομισματικές πολιτικές για τον κύριο Φερνάνδη πάντα, τη διασύνδεση δηλαδή τη δική μου έκθεση με την έκθεση του κύριου Τάγκ. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ω προ αυτό. Συνεργαζόμαστε και εγώ και ο κύριος ε, Τάγκ ε, με τους υπολείπους προς αυτό το σκοπό και σας ευχαριστώ και όλους εκ των προτέρων γι' αυτό. Για τη βελτίωση των κεφαλικών απαιτήσεων σε σχέση με μη είναι επικοδομητικέ προτάσει σα. Ήδη ο στόχο μα, κύριε Φερνάντε, ίσω να έχουμε απλά κάποιε διαφορετικέ απόψει, οπότε πρέπει να αναζητήσουμε συμβιβασμού. Έρχομαι στον κύριο Καμάλ. Κατανοώ τι ανησυχίε σα σε σχέση με την έργαση επαναλαμβάνω ότι ο στόχος νομίζω είναι κοινό και με κάποιες συμβιβαστικέ προτάσεις νομίζω θα καταφέρουμε να τον πετύχουμε. Επίσης συμφωνώ ότι πρέπει να μειωθεί η πολυπλοκότητα και συμφωνώ και εγώ ότι οι δύο, σχέσεις, οι δύο εκθέσεις, ε, ΤΑΝΚ και η δική μου, είναι συνδεδεμένες. Κύριο Στόιρερ, από τους φιλελευθέρους έκανε κάποιες εκτιμήσεις ε, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά τέτοιων προϊόντων ε, στη δέκα της κρίσης και συμφωνώ με την εκτίμησή του. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το στίγμα σε αυτά τα προϊόντα πλέον και θα πρέπει να είμαστε πολύ αποφασιστικοί και να προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε, να εκπαιδεύσουμε αν θέλετε, ε, ώστε να φύγει αυτό το στίγμα από αυτά τα προϊόντα σε ό,τι αφορά αυτά τα ABCP, τα Asset-Based Commercial Papers, τα χρεόγραφα που είναι καλυμμένα με περιουσιακά στοιχεία, τέτοιου είδους προϊόντα είπατε ότι δεν πρέπει όπως και ούτε και αξιολόγησης να επηρεάζουν αρνητικά την πραγματική οικονομία και συμφωνώ και εγώ. με την ανησυχία σας ό,τι αφορά τα σχόλια του κυρίου Ντεμάση από την ΚΟΕ αληθεύει ότι πρέπει να, είμαστε, ε, να έχουμε πείγνωση και να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε κάποιο συμβιβασμό για τον ρόλο των εικόνων αξιολόγηση. Καταλαβαίνω και κατανοώ την κριτική σας ή την ανησυχία σας αν θέλετε σε σχέση με την εσωτερική προσέγγιση, το internal approach. Σε ό,τι αφορά ε, κριτική που κάνετε στη μείωση των ελάχιστων απαιτήσεων σίγουρα είναι σημαντική η χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Υπάρχουν κάποιε αμφιβολίε για το αν αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Εγώ είμαι πεπισμένο προ αυτό, όμω είμαι ανοιχτό και σίγουρα θα έχουμε διάλογο στα θέματα αυτά. Ο κύριο Βάλλη λέει ότι δεν θα βοηθηθούν οι ΜΜΕ. Εγώ ελπίζω να βοηθηθούν. Αυτό είναι ένα κοινό μα στόχο. Εσεί έχετε άλλε προτάσει για τη βελτίωση της κατάστασης ε, για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ και είμαστε διατεθειμένοι να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ Παμπλό. Ολοκληρώνεται αυτό το σημείο. Θα ανακοινώσω και το εξή. Στις 20 Ιουλίου είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών για το STS εκθεσιτάν και 22 Ιουλίου 12 το μεσημέρι για την έκθεση Παύλο θα το ονομάσουμε έτσι θα ψηφορία στην Επιτροπή μας προβλέπεται το φθινόπωρο και τέλος του έτους ψηφοφορία στην Ολομέλεια σύντομη διακοπή για να έρθουν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Απασχόλησης και μετά θα έχουμε την κοινή συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ.